Αγαπητοί φίλοι, γνωρίζω ότι έπεσε χιόνι στις Βρυξέλλες, αλλά επειδή ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες έχουμε μια αρκετά φορτωμένη μερίσια διάταξη, θα σας πρότεινα να ξεκινήσουμε. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 11 ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης θα το συζητήσουμε πριν το σημείο 7. Θα το ψηφίσουμε μάλλον. Σημείο 2. Ε, μην κάνετε μορφασμούς όταν μιλάτε. Γιατί αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Οπότε όποιες γκριμάτσες κάνετε και μορφασμούς θα τις δουν οι θεατές. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρία 10 Ιουλίου, 6 Σεπτεμβρίου και 17-18 Σεπτεμβρίου. Αν μέχρι τέλο συνεδρία δεν υποβληθούν παρατηρήσει, τα πρακτικά μα θα θεωρηθούν ω εγκεκριμένα. Σημείο 4. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησής μας, τον κύριο Φιλίπ Μπούλον, ο οποίος ε, εκπώνησε γνωμοδότηση που θα επιδοθεί στην αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή την ΤΕΒΕ ε, με θέμα τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση υπερπόντια σύνδεση. Ε, πρόταση απόφαση του Συμβουλίου. Και ο κύριος Πατρίς Τυρολιά είναι ο εισηγητής της έκθεσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εμείς θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Μπουλάου, στον οποίο δίνω και το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως είπατε, θα πρέπει η Επιτροπή μας να εκπονήσει γνωμοδότηση, την οποία θα δώσει την αρμόδια επιτουσίας Επιτροπή, την Επιτροπή Ανάπτυξης, με θέμα τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και δαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι είναι οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη, η ΧΕ. Πρόκειται για νησιά που συνδέονται με τέσσερι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τι κάτω χώρε. Δεδομένη της γεωγραφικής θέση και του φυσικού του πλούτου, ενδιαφέρουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η φόρος του ανάπτυξη. Η, συμφωνία του 2001, η απόφαση για τη σύνδεση πρέπει να τροποποιηθεί δεδομένων των ε, νέων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και του διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει οι υπερπόντες χώρες και δάφη να φέρουν την οικονομία τους στον δρόμο της οηφόρος ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και μειώντας τον ευάλωτο χαρακτήρα τους, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον σε συνεργασία με τους γείτονες και με ένταξή τους στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και στις δράσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Κατέθεσα 41 τροπολογίες ζητώντας να αναλυφθούν δράσεις ε, για την ε, προώθηση και σεβασμό των ε, κοινωνικών προδιαγραφών και στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενισχύουμε τους ανθρώπινους πόρους με προγράμματα διαβίου κατάρτισης, επαγγελματική επιμόρφωσης και βελτίωση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση. Επίσης, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες θα τονώσει την καινοτομία και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Πρόσθεσα και ένα άρθρο με την τροπολογία μου 32 για την υγεία και την προστασία στην εργασία ώστε να εξυγχρονιστούν οι δράσεις και να μειωθεί ο κίνδυνος από εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι συντομία. Είναι τα θέματα που πραγματεύομαι στην γνωμοδότησή μου και ε, προσβλέπω συνεργασία με τους χιώδης συγγητές για την περαιτέρω επεξεργασία της. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κρυβητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ηγήτρια των σοσιαλιστών για το θέμα αυτό και θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να σας κάνω πολύ σύντομη παρουσίαση των θέσεών μου ως σκιώδης συγγήτριας. Όπως σας είπα, είμαι η σκιώδη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και πιστεύω ότι με πολύ πρόσφορες συνθήκες θα έχουμε αγαστή συνεργασία με τον συντάκτη της γνωμοδότης, τον κύριο Φιλίπ Μπουλόμ. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι έχω καταθέσει 12 τροπολογίες, τις οποίες προσπαθώ να εξηγήσω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των υπερπόνδιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή των βαλτιστών πρακτικών για την απασχόληση, για τον κοινωνικό διάλογο και ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Επίσης, ε, ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπερπόντες χώρες και οι διαμερίσματα θα πρέπει να συνεργάζονται για να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία στην ε, πρόσβαση στην αγορά εργασία, αλλά και στην ε, υγεία και ασφάλεια στην αγορά εργασία. Επίση, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή τη ευελιξία με ασφάλεια, ώστε να αποφύγουμε κατακαιρματισμό τη αγορά-εργασία και να ε, τον αντισταθμίσουμε με καλές κοινωνικέ συνθήκε. Επίσης θέλουμε συνεργασία για τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ε, για παρόχες ε, φροντίδας παιδιών, ε, βρέφων βρέφονιπιακού σταθμούς και επίσης να λάβουμε υπόψη και την ισότητα των δύο φύλων ή την, τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και φυσικά τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Ίσως κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι. Οπότε κύριε Μπουλό, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον όλα φαίνονται μια χαρά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν βέβαια. Θέλετε να απαντήσετε στη σκιώδη συγγήτρια. Όχι όντως, ε, φαίνεται ότι θα διεξαχθεί απρόσκοπτα η συνεργασία μας. Πολύ ωραία, η Ευρώπη προοδεύει. 14 Ιανουαρίου λίγη προθεσμία για τις ε, τροπολογίου, συγγνώμη, 11 Νοεμβρίου. Στις 14 ε, Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τι τροπολογίε ε, για να δούμε αν θα υποβληθούν στι 23 Ιανουαρίου συμβαστικέ τροπολογίε ώστε να ψηφίσουμε την επαύριο και 18-19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσει η αρμόδια Επιτροπή ΔΕΒΕ. Θέλουμε να προλάβουμε ώστε να δώσουμε γέρο στην γνωμοδότησή μα για να ληφθεί υπόψη. Για το σημείο 5 τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντία Μακεντάιρ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της με θέμα τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Η γνωμοδότηση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας του Ανδρέα Σβάπ. Κυρία Συγγέντρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς είχαμε ήδη μια σύντομη ευκαιρία να συντάξουμε κάτι για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και όλοι θεωρήσαμε ότι αξίζει τον κόπο να ακουστεί και η γνώμη της Επιτροπής Απασχολήσεως για λογαριασμό δηλαδή της ε, Επιτροπής Ενίας Αγοράς σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν απασχόληση. Πάλι εδώ, σε τούτην εδώ την γνωμοδότηση, λέμε ότι ανοίγονται μεγάλες ευκαιρίες με την ενιαία αγορά και υπάρχει βεβαίω η δυνατότητα <clears throat> πάντοτε οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις ιδίω εφόσον ε, λάβουν βοήθεια να ενισχυθούν Λέμε επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με απλούστευση διαδικασιών, με ευκολότερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Δηλαδή έχω προσπαθήσει να περιλάβω ένα σφάσμα διαφόρων ε, πραγμάτων. Βέβαια το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ ε, σφιχτό. Όχι επειδή εγώ το ζήτησα, αλλά όλα γίνονται στα αγγλικά. Θα έλεγα λοιπόν, εάν κανείς εκ των σκιωδών εισηγητών επιθυμεί να καταθέσει τροπολογίες. Πολύ ευχαρίστως να συνεργαστώ με τα πρόσωπα αυτά, ώστε να μπορέσουμε ή δυνατόν, ελπίζω, να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη γνωμοδότηση και να προωθήσουμε έτσι τη θέση της Επιτροπής μας με επικοδομητικό τρόπο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος κυρία Μπέρες. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του συναδέλφου Κοτσολίνο θα ήθελα να εκφράσω την γενική συμφωνία μας με την έκθεση McIntyre με, με μια μικρή επιφύλαξη. Ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι μικρό αλλά έχει αρκετή πολιτική σημασία. Στην παράγραφο 8 Η κυρία Μακιντάιρ ζητά να καταργηθούν ε, απαιτήσει νομοθετικές για την δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτό συνήθως συνδυάζεται με ένα αίτημα κάποιων πολιτικών ομάδων να περιοριστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και ιδιαίτερα ε, των υγειονομικών διατάξεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία προκειμένου να δοθούν ενάψματα για δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση κτλ. Κυρία Μακιντάιρ, νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίγνωση ότι είναι αρμόδια ε, και θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι κανόνες ασφάλειας, οι προδιαγραφές ε, υπέρ της προστασίας, της υγείας και της αξιοπρέπειας στην εργασία να υπερτερούν οποιασδήποτε άλλες ανησυχίες. Μπορεί άλλες ε, επιτροπές να ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει η δική μας επιτροπή να προσπαθεί να αποδυναμώσει την ήδη ε, χαλαρή νομοθεσία που έχουμε για τα θέματα αυτά γιατί έχουμε απλώς μια οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, με ελάχιστες προδιαγραφές. Δεν θα πρέπει και αυτές τις ελάχιστες προδιαγραφές να τις αποδυναμώσουμε περαιτέρω, να τις υποτιμήσουμε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με την παράγραφο 8. Και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία θα ζητήσουμε ίσως και διαγραφή της. Ευχαριστώ. Est-ce qu'il Υπάρχουν άλλα σχόλια. Ο κύριος Κόζας. Η κυρία Κόζας. Α, με συγχωρείτε. Ναι, Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να συντάξουμε την έκθεση, την γνωμοδότηση και έχουμε μόλις μία εβδομάδα για να καταθέσουμε τις τροπολογίες. Εγώ είμαι εισηγητής εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚΑ και χθες το κοίταξα λίγο και θα ήθελα να συγχαρώ ε, ε, να σας συγχαρώ γιατί παρά το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ε, έχετε φτιάξει μια πολύ περιεκτική και πυκνή γνωμοδότηση. Εάν υπάρξουν τροπολογίες από το ΕΛΚΑ εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους άλλους εισηγητές, τους εισηγητές και τον ε, αρμόδιο της ουσίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε όσο γίνεται πιο ομαλά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Η Κομισιόν είναι παρούσα, θέλει να παρέμβει. Όχι. Κυρία εισηγήτρια, θέλετε να κλείσετε. Όχι. Δεν είναι ναι, ναι, απαραίτητο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε προθεσμία κατάθεση προθεσμιών μόνο στα αγγλικά 11 ε, ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Ε, ε, Δεκεμβρίου με συγχωρείτε. Ε, και 18 Δεκεμβρίου θα ξαναεξετάσουμε τις τροπολογίες που θα είναι στα αγγλικά και θα τις ψηφίσουμε την ίδια μέρα, 14 πρώτου. Ούτως ώστε η Επιτροπή και Αγορά να μπορέσει να τις λάβει υπόψη στην ψηφοφορία 23 και 24 Ιανουαρίου. Και περνάμε στο σημείο 6. Comme vous le savez, là, euh... Όπου έχουμε μάλλον πρέπει εγώ να σας παρουσιάσω μετά από αίτημα των συντονιστών ένα σχέδιο προφορικής ερώτησης και δύο ψηφίσματα για την εγγύηση των νέων. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έθεσε επιτάπητος υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Αντόρα ένα σχέδιο εγγύησης νέων όπως είναι και η πρόταση, σύμφωνα με την πρόταση μάλλον προέκυψε από την Κομισιόν, στην ουσία πρόκειται για μια πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν στο μέτρο του δυνατού το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να κάνουν τέτοιες εγγυήσεις νέων, δηλαδή δεν είναι ευρωπαϊκός ε, οργανισμός, αλλά είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός που σέβεται απολύτως τις αρχές της επικουρικότητας. Και παραλλήλως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης της ανάπτυξης υπέδειξε ότι αυτή η εγγύηση νέων θα μπορούσε να συνδυαστεί με το πλαίσιο των όσων γίνονται μέσα στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και σύγκλησης των κρατών μελών και άρα να χρησιμοποιηθεί στις ε, συστάσεις προς κάθε χώρα. Το εν λόγω σχέδιο λοιπόν και το σχέδιο ψηφίσματος που έχετε μπροστά σας, στόχο έχει, πέρα από τις επιτυσσουσίες εργασίες που θα γίνουν και που είναι ευθύνη των εισηγητών που έχουμε ορίσει στο πλαίσιο μιας έκθεσης πρωτοβουλίας και μιας ε, συσχέτισης με τις εργασίες της Επιτροπής ε, Πολιτισμού Επιθυμία λοιπόν των συντονιστών ήταν να έχουμε μια ειδοποίηση ή εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερη ορατότητα του Ευρωκοινοβουλίου πριν ε, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ της 16 Φεβρουαρίου να λάβει θέση επί αυτής της σοφής και ταπεινής ε, σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο που έχετε λοιπόν συντάχθηκε πριν να έχουμε το κείμενο της και γι' αυτό θα ήθελα να σας προτείνω στο ίδιο το τα άρθρα του, του ψηφίσματος να προσθέσουμε ίσως μια-δυο παραγράφους πιο συντονισμένες με τα όσα μας υπέβαλε η Επιτροπή, διότι στην πράξη τα ισχυρά σημεία είναι αυτά που είπαμε, το έφεση και η χώρα συστάσεις. Δεν είναι και τίποτα το εξαιρετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έχουμε να μελετήσουμε ως πρόταση. Εάν λοιπόν αυτό τελικά θα περάσει, θα πρέπει να πούμε κάτι και ζητώ συγγνώμη που δεν το έχω ήδη συντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι που να λέει είναι της άποψης ότι αν αυτή είναι η σύσταση που δέχονται τα κράτη-μέλη. Και όπως σας είπα δεν το έχω συντάξει, το λέω έτσι τώρα προφορικά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι συνεπή και να επιτρέψουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέχρι 25% στις πολιτικές Ε, να προβλέψουν δηλαδή ένα κονδύλι στην πολιτική συνοχή που θα επιτρέπει ε, να χρηματοδοτείται αυτό το νέο ε, αίτημα που βαραίνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και αυτή είναι η πρώτη συμπληρωματική πρόταση και η δεύτερη είναι να ξαναπούμε πόσο πολύ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη να ενσωματώσει αυτή τη διάσταση στις συστάσεις τη στιγμή που θα συντάξει τις αναχώρα συστάσεις. Ξέρω πως το αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος δεν είναι να σας πούμε τι θα κάνουμε ε, στη συνέχεια, αλλά εφόσον θέλουμε να επηρεάσουμε, πρέπει να επηρεάσουμε πριν το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Προσθέτοντας δύο στοιχεία αυτά που σας ανέφερα και ζητώ και πάλι συγγνώμη που δεν τα έχω συντάξει η κυρία Ρολάν και μετά ο κύριος Κρίστενσον και η κυρία Ρολάν Σαρτιέ. Πριν σας δώσω το λόγο να σας προτείνω ότι όταν θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος απόψε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, χωρίς να γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα, να ενσωματώσουμε αυτό το σημείο γιατί αυτό το σημείο είναι νέο. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ανάμεσα στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και το διάλογο του για το κοινωνικό ταμείο, δεν τα πρόσεξα όλα. Και άρα μόλις τώρα βλέπω αυτό το προφορικό ερώτημα και το σχέδιο ψηφίσματος. με το οποίο βασικά συμφωνώ. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι συμμετέχω στον τριμερή διάλογο και ξέρετε πως ε, σήμερα το απόγευμα θα σας βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, έχω την εντύπωση και αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά σκληρής συζήτησης στο Συμβούλιο στον τριμερή διάλογο την περασμένη εβδομάδα τελευταία δηλαδή επαφή που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι δηλαδή πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε πιο ταπεινοί, πιο ανοιχτοί και πιο ε, δραστήριοι. Κά Υπάρχει κάτι όταν μελετάμε την κατάσταση των νέων 18 με 25 ετών που έχουν δυσκολίες να μπουν στην αγορά εργασίας και αν αυτά τα διασταυρώσουμε με τα χαρακτηριστικά της εξόδου από, χωρίς ε, δεξιότητες, χωρίς, χωρίς διπλώματα, Νομίζω ότι εάν προτείνουμε κάτι θα πρέπει να προτείνουμε την επιστροφή στην κατάρτιση γιατί πολύ συχνά αυτοί οι νέοι βγαίνουν από συστήματα κατάρτισης και θα πρέπει να αναφέρουμε και μια, μια, άλλη οδό που είναι τα προγράμματα κινητικότητας, τα προγράμματα εθελοντισμού, τα... και για αυτούς τους νέους που δεν είναι ενσωματωμένοι στα συστήματα κατάρτισης, πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να τις αναφέρουμε αυτές τις δυνατότητες, γιατί διαφορετικά απέτυχαν μια φορά, θα επανέλθουν, θα, αποτύχουν και πάλι και ίσως και να έχουν ε, πολλές φορές αποτύχει. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με άλλα προγράμματα, να τους κινητοποιήσουμε με τα προγράμματα κινητικότητας, εθελοντισμού και να συμπληρώσουμε άρα τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν για τους νέους. Γιατί είναι αποτελεσματικές αυτές οι πολιτικές. Και γι' αυτό το λόγο και στις, στις εθνικές πολιτικές καταπολέμησης της εξόδου των νέων από το σύστημα παιδείας άνευ προσόντων θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να φτιάξουν μια πορεία προσωπική. Έχουμε μακροσκελή κατάλογο ομιλητών. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αντικείμενο της προφορικής ερώτησης και του ψηφίσματος δεν είναι η ανάλυση όλου του θέματος της εγγύησης για την νεολαία. Γιατί έχουμε σχετική έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Της κυρίας Ξιντλεύσκα και εντάσσεται αυτό στι κοινοβουλευτικέ μα εργασίε. Θέλουμε απλώ να στείλουμε ένα μήνυμα με την προφορική ερώτηση με βάση την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ε, του Φεβρουαρίου. Ε, παρακαλώ σύντομα. Ναι, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπράξει το λάθο το ξεχάσει αυτό, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εμεί μπορούμε να το διορθώσουμε. Όλε Κρίστερσεν και μετά ενάντια Χίρσου και σας θέρμο παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρέπει να προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Ένα μεγάλο μέρος του Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να αφιερωθεί σε επενδύσεις, διότι αυτή τη στιγμή χάνουμε τον έλεγχο της ανεργίας των νέων δεν μπορούμε να αρκούμαστε πια σε λόγια. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το βάρος που έχουμε ρίξει μέχρι τώρα σε περικοπές, σε δημοσιονομικές περικοπές, σε περικοπές των δαπανών, έχει οδηγήσει σε τεράστια ενεργεία των νερών. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις, τεράστιες επενδύσεις. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιήσει κονδύλια, αλλά και οι χώρες μέλη. Αλλιώς ποτέ δεν θα ξεπεραστεί η κατάσταση αυτή. Γνωρίζουμε ότι στην Ισπανία η κατάσταση είναι τραγική. Το ίδιο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε οι νέοι άνθρωποι να είναι αυτοί που τελικά πληρώνουν το λογαριασμό. Χάνουν. Να διαχείρισω και μετά Αλεχάνδρος Σέρκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η πρωτοβουλία για τις εγγυήσεις υπέρ των νέων είναι πολύ σημαντική. Πρέπει ταυτόχρονα να είναι σαφές ότι με αυτή την εγγύηση υπέρ των νέων δεν δημιουργούμε απασχόληση. Την απασχόληση θα δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που σημαίνει δηλαδή αυτή η εγγύηση είναι ότι προσφέρουμε μια δυνατότητα μετάβασης μέχρι ότου βελτιωθεί η κατάσταση. Ασφαλώς μετά έχει νόημα να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του κοινωνικού ταμείου, να δούμε πώς μπορούν να αποκτήσουν οι νέοι περισσότερα προσόντα, ειδικά η ομάδα εκείνη των νέων που λόγω ελλείψεως προσόντων βρίσκεται σε ούτως ή άλλως μειονεκτική κατάσταση. Αυτά πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερως. Γιατί εγώ βλέπω ότι αυτή η ιδέα της Youth Guarantee έχει μεν θετική απήχηση, αλλά χθε άρχισαν να την συνδυάζουν τουλάχιστον τα γερμανικά μέσα με μια job guarantee, δηλαδή με μια εγγύηση ότι θα βρουν δουλειά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Να μην ξυπνήσουμε κάποιες προσδοκίες που ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε γιατί αυτό που αποσκοπεί εδώ το μέτρο αυτό είναι να δώσει τη δυνατότητα μιας μεταβατικής περίοδου για τους νέους. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο Αλεχάνδρος Σέρκας. Και μετά κύριε Κορνέλησε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι και εμείς εστερνιζόμαστε τη γνώμη σας ότι θέλουμε μια νέα παράγραφο στο ψήφισμα όπου θα προσδιορίζουμε τη θέση μας μετά την έγκριση αυτής της πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα μικρό σχόλιο. Διάβασα και τη σχετική τεκμηρίωση και τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως είπατε, επαφείται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Από αυτά εξαρτάται τι θα γίνει. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική δημοσιονομική ευρωπαϊκή δέσμευση. Εξαρτώνται τα πάντα από τα κράτη-μέλη. Οπότε αν προσθέσουμε εμείς μία παράγραφο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και 7 χρόνια τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα. Από τις κατευθυντήριες γραμμές ε, του 2005 ακούγαμε αυτό το θέμα της εγγύησης για την νεολαία, αλλά τίποτα δεν έγινε και δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό το κοινωνικό ταμείο. Από το 2005 το ακούμε λοιπόν και μέχρι στιγμής τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Θα Πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να γίνει πραγματικά μια ευρωπαϊκή εγγύηση για την νεολαία, να μην είναι μια γραφειοκρατική απλώ διατύπωση. Να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αλλιώ που δεν είδα θα πρόκειται για ευρωπαϊκή εγγύηση για την νεολαία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Εμίλιο Τουράναν που δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Εμένα με ικανοποιεί και η προφορική ερώτηση και το κείμενο του ψηφίσματος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επιτέλους το πακέτο για την νεολαία. Είναι από τις ελάχιστες φορές ε, στην κοινοβουλευτική μας θητεία που μια έκθεση πρωτοβουλίας πραγματικά προκάλεσε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εισακούστηκε από αυτήν η επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σπάνιο πράγμα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Γι' αυτό και υποστηρίζω αμέριστα αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια, οι χώρες που περισσότερο χρειάζονται τέτοιες δράσεις δεν έχουν κονδύλια για την εγγύηση των νέων. Χρειαζόμαστε και εδώ περισσότερη αλληλεγγύη και αυτό φαίνεται στην προφορική ερώτηση. Φυσικά θα συνεργαστεί ο κ. και με τους και ηγητές και είναι υπέρ της ε, προσθήκης των δύο παραγράφων που πρότεινε η πρόεδρος, αλλά θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Κυρία Στανλού και μετά κυρία Μακιντάιρ. Σας ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία είναι θετική και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιο μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Στόχος της Youth Guarantee πρέπει να είναι να ενταχθούν οι νέοι στην πρώτη δουλειά στην πρώτη αγορά εργασία. Τα προγράμματα κινητικότητα μπορούν να παίξουν ρόλο συμπληρωματικό. Δεν λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Επίσης τα προγράμματα των εθελοντών βάζουν τους νέους σε κάποια δραστηριότητα, δίνουν κάποια προσόντα, αλλά όχι απαραίτητα θέση δουλειάς στην πρώτη αγορά εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει δεσμευτικά να αναθέσει στις χώρες μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να τους επιβάλλει βέλτιστες πρακτικές όπως έχουμε κάνει και για την καινοτομία και αλλού, ώστε και να ανταλλάσσονται καλά παραδείγματα, αλλά και είμαι και πεπισμένη ότι μετά από τόσα χρόνια εθελοντικών ε, πρωτοβουλειών στην ε, ανεργία των νέων, για, κατά της ανεργίας των νέων δηλαδή, δεν έχουμε προχωρήσει. Η Youth Guarantee είναι σημαντική και για την απόκτηση προσόντων. Μας λένε συχνά οι επιχειρήσεις ότι δεν έχουμε καλά εκπαιδευμένους νέους. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που αν ληφθεί υπόψη σοβαρά, αν δηλαδή εκτελεστεί σοβαρά, θα μπορέσει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων των νέων. Καθώς επίσης να αντιμετωπίσει και την έλλειψη των ειδικευμένων εργατικών χεριών. Άκουσα και από την βιομηχανία πάντως και στη Γερμανία ότι η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται θετικά. Μακιντάιρ. Ευχαριστώ. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε και όλες ότι η ανεργία των νέων είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτή εδώ η εγγύηση νεολαίας. Όντως ε, θα λύσει τα πραγματικά προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να ακουστούν δηλώσεις που ηχούν ωραία, αλλά να μην γίνει τίποτα. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Εάν ε, μάλλον δεν είναι οι κυβερνήσει. ούτε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα δημιουργήσουν δουλειέ. Οι επιχειρήσει θα δημιουργήσουν δουλειέ. Δεν μπορεί να νομοθετήσει ότι θα δημιουργήσει απασχόληση. Ούτε θα νομοθετήσεις, ούτε μπορεί να νομοθετήσει ότι οι επιχειρήσει θα προσλαμβάνουν περισσότερου ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να βοηθήσει του νέου προσφέροντα εκπαίδευση και δεν πρέπει να αποδυναμωθεί το Κοινωνικό Ταμείο ούτε να κατασπαρούν οι δυνάμεις του. Γι' αυτό εγώ δίνω ιδιαίτερο βάρος εδώ στην ιδέα να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες του Ταμείου στην εκπαίδευση των νέων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας που προκαλούνται από το ότι δεν ταιριάζουν θέσεις με τα υπάρχοντα προσόντα. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ακαμψία στην αγορά εργασία. Με ανισχύει πολύ ότι θα προκαλέσουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη 15 λεπτά καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλη τη συζήτηση τώρα για την απασχόληση των νέων. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε πριν από το ΕΨΚΟ του Φεβρουαρίου. Έχω λοιπόν ακόμα τρεις εγγεγραμμένους να είναι πολύ σύντομοι και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφόρια. Ορί, Σανκλέρ, Σλοβιέτσκα και εδώ κλείνει ο κατάλογος των αγορητών. Ορί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την εγγύηση των νέων και είναι ένα θέμα ιδιαίτερο προσφυλές για μας θέμα αλλά είναι βέβαια η χρηματοδότηση Μιλάμε βέβαια για το κοινωνικό ταμείο όντω, Αλλά θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις ε, προτάσεις και για το Ταμείο Συνοχής και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής. Γιατί έχουμε μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πολλές χώρες. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες θα καλύψουν αυτή την εγγύηση για την νεολαία. Ευχαριστώ. Η κυρία Σενκλέρ, η κυρία Γιαζοβιέσκα και τελειώσαμε με τους ομιλητές. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να επανέλθουμε στο θέμα. κυρία Σενκλέρ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Η ενεργεια των νέων είναι μάστιγα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στη δική μου εκλογική περιφέρεια, τα West Midlands. Και η πρωτοβουλία αυτή, παρόλο που είναι καλοπροαίρετη και περιλαμβάνει πολλέ βαρύγδουπε δηλώσει και ωραία λόγια, δεν νομίζω ότι θα φέρει λύση. Το θέμα δεν είναι να ε, ε, επιβάλλουμε υπερβολικέ ρυθμίσει ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που εξασφαλίζουν 83% των θέσεων απασχόληση. Γιατί η υπερβολική νομοθεσία επιβαρύνει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε αν θέλετε όντως να δημιουργήσετε ε, θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο, στη Μεγάλη Βρετανία, να σταματήσετε τις υπερβολικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρία Γεωζοβέσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για την κατάρτιση, την επιμόρφωση, για τις εγγυήσει ε, στην εργασία για τους νέους και Μιλούμε πολλές φορές ε, για τους νέους που είναι οι αποδέκτες αυτών των προτάσεων, αλλά δυστυχώς όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι, οι θέσει απασχόληση δεν δημιουργούνται ούτε από την κοινωνία ούτε από το κράτος, αλλά από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιου μηχανισμούς ε, και κάποιε εγγύησει ώστε να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι που δημιουργούν τι θέσει εργασία. Και επίση να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα των νέων. Γιατί χρόνια ολόκληρα μιλούμε για τι εγγύσει για την νεολαία και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο πάντα. Έχουμε δυστυχώ ένα μεγάλο αριθμό νέων, 18 με 25 ετών, που ούτε σπουδάζουν, ούτε παρακολουθούν κάποια κατάρτιση, ούτε εργάζονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των νέων είτε στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, είτε σε, διάφορες, σε διάφορα στάζ, σε μαθητείες είναι σημαντικό ε, να ενισχύσουμε έτσι την επιχειρηματικότητα των νέων για να μπορέσουν και οι ίδιοι να ξεκινήσουν ενδεχομένω και μια δική του ε, επαγγελματική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά του συναδέλφου. Βλέπουμε ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και είναι σημαντικό η Επιτροπή μα Κοινωνικών Υποθέσεων και απασχόληση ε, να ενεργοποιηθεί για το θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα λοιπόν να μακρηγορήσω γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίε μας αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε ένα σχόλιο που άκουσε επανειλημμένος, ότι δεν θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί το νομοθετικό, το κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να ευνοήσει ή αντίθετα να παρακολύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό διακύβευμα και με αυτό ασχολούμαστε και εμείς ώστε να αποτρέψουμε μια τέτοια παρεμπόδιση. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα, το αντίθετο. Αλλά από τις εμπειρίες που έχουμε σε πολλά κράτη-μέλη, στην Αυστρία, στη Φιλανδία, στο Λουξεμβούργο και στη δική μου την πατρίδα, τη Γαλλίδα, όπου οι συμβάσεις ε, μεταξύ των γενεών ε, είναι πρωτοβουλία και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι μηνύματα ότι και οι κρατικές αρχές, οι δημόσιες αρχές μπορούν να αναλάβουν δράση προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διαβιβάσουμε το μήνυμά μας στο Συμβούλιο και να πούμε μέσω του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και σαφέστατο μήνυμα εγώ θα είμαι η εκπρόσωπό σας στο φερέφωνο σα σε αυτό το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων ε, και Απασχόλησης ε, τη 17 Φεβρουαρίου, που θα είναι άτυπο και έχω λάβει ήδη από την Ελλανδική Προεδρία τη σχετική πρόσκληση. Οπότε δείξτε μου εμπιστοσύνη, θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα και μάλιστα μεταφρασμένο στη Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Τώρα, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι συντονιστές ε, θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να καταθέσουν τις τροπολογίες τους στα αγγλικά και σας ζητώ συγγνώμη που επιβαρύνω εδώ τους συντονιστές και θα ήθελα αυτή να αναλάβω το θέμα. Λοιπόν, τροπολογίες στα αγγλικά υπό την αιγύδα και την ευθύνη των συντονιστών 11 Δεκεμβρίου το μεσημέρι λίγη προθεσμία ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε ήδη από τις 18 Δεκεμβρίου τις τροπολογίες. παραλαμβάνω, δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση εφόλης της ύλη για το θέμα των νέων. Απλώς θα στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Γι' αυτό και το, σύντομο, το ψήφισμά μας θα πρέπει να είναι σύντομο. Γιατί φαντάζεστε ότι όσο πιο μακροσκελές είναι το ψήφισμα, ε, τόσο πιο δύσκολα θα γίνει κατανοητό ή θα προκαλέσει την προσοχή. ξεπερνάει τη σελίδα, ούτε πρόκειται να ρίξουν καμιά ματιά οι υπουργοί. Θα πρέπει να είναι συνοπτικό και μεστό. Τώρα, για το σημείο 11, σας έχει υποβληθεί ένα σχέδιο εκθεσής με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Όπως ε, θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, δεν έχουν αλλάξει οι περιστάσεις και οι συνθήκες απασχόλησης στα κρατημέλη και ούτε οι κατευθυντήρες γραμμές έχουν αλλάξει. Οπότε τις παραπέμπουμε όπως τις εγκρίναμε αυτούσιες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μετά την έκθεση όρη. Μπορείτε να δέχετε λοιπόν την, ε, το σχέδιο έκθεση όπως έχει υποβληθεί. χωρίς αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, τυπική διαδικασία. Και σας ζητώ συγγνώμη για την γοητεία αυτή της τυπικότητας. Λοιπόν, προχωράμε στις ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση κυρίας Ρεζίνα Μπάστος. Έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ελληλασφάλισης. Ε, εδώ ισχύει η διαδικασία ε, συνεργασίας μεταξύ επιτροπών. Έχουμε κοινή αρμοδιότητα με την ε, νομική επιτροπή. Έχουμε συμβαστική τροπολογία, ένα α. Διακόπτη πρόεδρος. Μου διέφυγε το αστείο, εν πάση περιπτώσει. Ίσως κάποιος έχει την καλοσύνη να μου εξηγήσει αργότερα. Παράγραφος 1 Τροπολογία Μπεναμιά. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Κυρία Μωράν Σαρτιέ, η συγκίτρια ίδια είναι υπέρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κυρία Μωράν Σαρτιέ, συγγνώμη. Αλλά εγώ δεν έχω πάρει το κατάλογο ψηφοφόρη. Και δεν είμαι η μόνη. Ολόκληρη ομάδα μου δεν έχει λάβει. Εντάξει, ευχαριστώ. Το ΕΛΚ φαντάζομαι συμφωνεί με την εισηγήτρια την κυρία Μπάστος. Δεν θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά σας. Λοιπόν, τροπολογία 2. Την αφήνουμε για αργότερα. Μετά την παράγραφο 1 ψηφίζουμε τη συμβεστική τροπολογία Α από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 καταπίπτει. Και μετά την τροπολογία 1, τροπολογία 4, Σίπελ, η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. Στην παράγραφο 2, η, παράγραφ, η τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 6 του κυρίου Ζανλίκ Μπεναμιάση. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 4, τροπολογία 7 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Για την παράγραφο 5, συμβαστική τροπολογία Β από τρει ομάδε, ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Καταπίπτουν σχετικέ τροπολογίε. Μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 11, μπάστο, ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5 και πάλι τροπολογία 12, χάρκι, ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Για την παράγραφο 6, συμβαστική τροπολογία σε τριών ομάδων, ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6, τροπολογία 15, Μαρά Σαρτιέ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16 τη ιδέα υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία 16 εγκρίνεται. Για την παράγραφο 7 τώρα, τροπολογία 17 έχει αποσυρθεί. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 18, Howitt, Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19, συμβατή, Ποιο είναι υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα από τρεις ομάδες υπέρ, κατά αποχέ. εγκρίνεται. Μετά την παραγραφή 8, τροπολογία 23, Σύπελ. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9 έχουμε την παράγραφο 24 κλειβέτη με προφορική τροπολογία της συγγετρίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 10, τροπολογία 25, Μωράν Σαρτιέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 σύπελ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 σύπελ συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 11 29 το κύριο Χόουιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Κλειβέτη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Μπεναμιάς. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 12. 33. Καταπίπτει. Παράγραφος 13. Τροπολογία 34. Σίπελ. Με προφορική τροπολογία της κυρίας ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Σίπελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν έχω την κάρτα μαζί. Tout le monde a Ψηφίσατε όλοι. Enfoncez bien vos cartes. Ah ben, si c'est la ligne des dirigeants qui ne marche pas. Bon, alors vous allez nous indiquer vos voix, vos, vos votes. Vous votez. Πείτε μας πώς ψηφίσατε τουλάχιστον. Ο κύριος Σωρία απέχει. Δύο υπέρ και δύο κατά. Λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 αργότερα. 37. Μπάστο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Μετά τη 14, τροπολογία 38, Χόουιτ. Ποιος είναι υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40, Μπεναμιάς, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39, συμβατή, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το 15. 41 Χόουιτ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 Κλειβέτη. Μινοδόρα κλειβέτη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 Σίπελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 Μπεναμιάς οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το κείμενο χωρίς τις φράσεις in και point out that διαφυλάσσοντας το, κοινωνικό, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Quarante-deux, 42, 26 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μό 45. 45 της ηγήτρια συμβατή ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 σίπελ μετά την παράγραφο 16 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 της ίδιας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 17, 48 Μαριάν Χάρκιν υπέρ. Ο παράγραφος 17, amendement 48. και Υπέρ, κατά τη 48 μιλάμε, αποχές εγκρίνεται. 49 συμβατή ψηφίζουμε, Σίπελ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συστάσεις τώρα. Μετά την παράγραφο 17, πρώτη σύσταση, ε συμβαστική λύση, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη σύσταση της κυρίας Μπάστος, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Για τη σύσταση 3, Έχουμε προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την 52 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεστική, ε, σύσταση, συγγνώμη, 4. Ησυχία παρακαλώ για να ακούγεται η φωνή μου. Πού είναι το σφυρί μου. Δεν έχω σφυρί. 53 μπάστο. Σύσταση 4 με προφορική τροπολογία της ίδιας εισηγητρίας. Ψηφίζουμε Ποιο είναι υπέρ τη 53. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την σύσταση 5 συμβαστική τροπολογία F από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F ήταν αυτή. Και φτάνουμε στην σύσταση 7, τροπολογία 56 ΣΥΠΕΛ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 56. Euh, Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 17 ψήφισαν υπέρ και 24 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 57 σύπελ υπέρ. Κατά. Νομίζω με την ίδια διαφορά, ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για την 57. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. 23 υπέρ, 24 λέει πρόεδρος υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 58 είπε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται λέει πρόεδρος. Α, συγγνώμη, λάθος, λάθος. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Heureusement Ψηφίζουμε το, το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί της έκθεσης ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Madame Bastos, je ne peux que vous inviter à Κυρία Μπάστος, αφού ολοκληρωθούν τα συγχαρητήρια του ΕΛΚ, θα ήθελα να σας πω εκ μέρους της Επιτροπής μας ότι μας ενδιαφέρει να είστε παρούσες στις διαπραγματεύσεις με την Νομική Επιτροπή, γιατί έχουμε εδώ κοινή αρμοδιότητα και παρακαλώ να με ερημνήσετε όταν γίνονται συναντήσει των σχεδόν εισηγητών στην νομική επιτροπή να λαμβάνονται υπόψη και οι δικέ μα απόψει. Όχι να οριστικοποιηθεί η δική του έκθεση ερήμην των δικών μα παρατηρήσεων. Αυτό ισχύει και για άλλα θέματα, αλλά παρακαλώ να το φροντίσει αυτό η συγκεκριά μας, να εισακουστούν τα αιτήματά μας στη Νομική Επιτροπή. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κάμπρνοχ, σημείο 8 της της διάταξης με θέμα την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γύρανση. Alors, euh, au paragraphe 1, nous sommes saisis d'un amendement de compromis A présenté par quatre groupes. Qui est pour Την παράγραφο 1 από 4 τροπολογίε συμβαστική υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 τις ίδιες ηγήτρες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 συμβαστική βήτα. Υπέρ κα, κατά αποχές εγκρίνεται. Qui est insupportable. Παρακαλώ, πάψτε να ψιθυρίζετε εδώ, δίπλα, στους διαδρόμους. Τροπολογία 10, Κέσλερ. Με προφορική τροπολογία δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11, κόντς, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12, Κάσλερ που θα μετακινηθεί αν εγκριθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Συμβιβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 19, ε, ε συμβαστική D, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 3, τροπολογία 24, μηνοδόρα κτιβέτη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 πέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Όχι, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 25. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 20 κατά. Μία αποχή έχετε δίκιο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Κίνκα Κούντζι Πέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Πέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 κίνκα Κούντζι Πέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 31 της κυρίας Γιακονσάρη. Για διαγραφή. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική ε που έχουν υποβάλει τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 36, Κίνγκα Κούντς, υπέρ, κατά, Οποχέ. Εγκρίνεται, 36 ε, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 37, Κάσλερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, συμβαστική F, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5 περνάμε στην 45, 47 Κάσλερ υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 47 για να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. 17 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. 48 Κίνγκα Κόντς υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 49 κλειβέτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 κούντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 5 52 καταπίπτει και έχουμε την παράγραφο 6 συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 της Αντιπροέδρου Ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 θα επαλχεύσουμε την 63 ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίζετε όλοι 24 υπέρ 16 κατά μία αποχή εγκρίνεται 64 κόντς υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Ρομπέρτα Αντζελίλη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Μαριάν Χαρκίν. Στη παράγραφο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 Αντζελίλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 Κίνγκα Κόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 ε, ε, Κάσλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 κόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 κόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά Του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 Ακολουθεί η τελευταία ψηφοφόρια του σημερινού πρωινού στο υπαριθμό 9 της ημερησίας διατάξεως έκθεση στα πλαίσια της συναπόφασης της κυρίας Μόραν Σοατιέ επί προτάσεως οδηγίας, τροποποίησεως δηλαδή, για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρομαγνητικά πεδία και άλλα σχετικά. Επομένως, γνωμοδότηση. Έχουμε γνωμοδότηση. Η κυρία Ράπτη επιθυμεί να λάβει το λόγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Κυρία Ράπτη. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να συγχαρώ από καρδιάς την εισηγήτρια Ελίζαμπεθ Μωρίν Σαρτιέ έκανε μια εξαιρετική δουλειά, μια δουλειά που απαιτούσε πολύ κόπο, πολύ υπομονή και πολύ ψυχραιμία. Θέλω να τονίσω και να επαναλάβω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος και τεχνικός φάκελος. Ε, έχουμε αγωνία για αυτόν το φάκελο όλοι μας, όχι μόνο εγώ ή η κυρία Σαρτιέ, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου με τους οποίους α, συζητώ συνεχώς και γι' αυτό ακριβώς ε, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις οι οποίες κατέληξαν χθες ε, παρακαλώ, εάν είναι δυνατόν, να υποβάλω μια προφορική τροπολογία στην αρχή του άρθρου 3, παράγραφος 2, η οποία τροπολογία δεν αλλάζει την ουσία του άρθρου που αφορά τις εξαιρέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό άρθρο, αλλά υπενθυμίζει κάτι που συνεχώς συναντούμε στα νομοθετικά κείμενα, την γενική αρχή του να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Καταλήγω λέγοντας ακριβώς στα αγγλικά για να διευκολύνω την πρόταση η οποία προτείνω να μπει στην αρχή notwithstanding the general principle of workers. Τηρείται ωστόσο η γενική αρχή ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εκτίθεται σε τιμές άνω των επιτρεπωμένων. Κλείνω λέγοντας το εξής. Ε, έχουμε δεχτεί όλες τις συμβιβαστικές και πραγματικά θέλω πάρα πάρα πολύ αν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία, ώστε αυτή η πολύ σημαντική έκθεση, αλλά και η πάρα πολύ σημαντική και καλή, εξαιρετική δουλειά της κυρίας Σαρτιέ, να συγκεντρώσει την υποστήριξη όλων μας. Εάν γίνει δεκτή η τροπολογία, υπερψηφίζουμε την, Amendment M. Εάν δεν γίνει δεκτή θα ψηφίσουμε αποχή. Και τελειώνω κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή. Ε, εάν δεν γίνει δεκτή σήμερα, δεν μπορέσουμε να την κάνουμε δεκτή σήμερα, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και πάλι και για μία ακόμη φορά ευχαριστώ την εισηγήτρια. Δεν ε, διαπραγματευόμαστε πλέον τώρα. Είμαστε λοιπόν στη συμβαστική M στο άρθρο 3 παράγραφος 2 όπου επιθυμείτε να προσθέσετε. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ακριβώ, ίσως η εισηγήτρια να άκουσε καθαρά το κείμενο. Αν θέλετε να το επαναλάβετε, μόνο την προφορική τροπολογία. Είναι κρίμα που δεν την υποβάλατε γραπτός, διότι αν την είχατε υποβάλει γραπτός θα είχε διανεμηθεί σε όλους. Έχετε δίκιο, λέει η κυρία Ράπτη, και ζητώ συγγνώμη. Και θα επαναλάβω την τροπολογία. Διακόπτη η Πού μπαίνει, πού μπαίνει στο κείμενο της συμβαστικής οι χώρες μέλη States shall require that the employers ensure that exposure, of workers, etc. Is, in είναι σελίδα 14 στις amendments, είναι η amendment M, το δεύτερο σημείο. Πριν από το δεύτερο σημείο που αρχίζει Member States shall require that the employers ensure, etc. Προτείνουμε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 the general principle of workers not being exposed above the exposure limit values. And then, member states... Okay, okay, okay. okay. Madame la Présidente, je... Ευχαριστώ την κυρία Ράπτη για τα λόγια της αυτά. Πάντως εμείς είμαστε αντίθετοι με την προφορική τροπολογία. Πρόκειται εδώ για μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Δεν μπορούμε την τελευταία στιγμή να δεχθούμε την προφορική αυτή τροπολογία. Καλώς, λέει η Πρόεδρος. Ερχόμαστε τώρα στη λίστα ψηφοφορίας. Άρθρο 1. Συμβιβαστική ζή. Έχουν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2. Συμβαστική ΚΑΠΑ. Πέντε ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3. Επί του τίτλου. Συμβαστική L. Πέντε ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Άρθρο 3. Η περίφημη συμβαστική M. Υπέρ. Την οποία υποβάλλουν τέσσερις ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Άρθρο 4. Επί του τίτλου ψηφίζουμε την 92 της κυρίας Ντελή. Η εισηγείται υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4. Συμβαστική N. 5 ομάδων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5. Συμβαστική όμικρον. 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6. Συμβαστική π. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8. Συμβαστική Q. 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 9. 178 του κυρίου Μαν η εισηγήτρια είναι αντίθετη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το άρθρο 9, νέος τίτλος, μεσοπροφορικής τροπολογίας της εισηγητρίας. Υπάρχουν ενστάσεις κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Τίθεται σε ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 9, 245 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί στο άρθρο 3 παράγραφος 5 νέα υποπαράγραφος α, εκπίπτει μετά το άρθρο 9 248 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 249 και σατχέ υπέρ κατά αποχές εγκρι... εγκρίνεται όντως άρθρο 10 συμβαστική ρο 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 11 παράγραφος 2 15 της κυρίας Σάτιε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 12 παράγραφος 1 τροπολογία 16 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 13 συμβαστική S 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 14 συμβαστική TAF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράρτημα 1. Συμβαστική ου. Πέντε ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Στο παράρτημα 2. Συμβαστική β. Πέντε ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 15, παράτημα 3, συμβαστική W, 5 ομάδων υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, παράτημα 4, συμβαστική X, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 5, 234 της Κεσουατιέ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ε, ε, το 6 συμβαστική α υπερ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Αιτιολογική σκέψη 7. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική 10. Σι 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική 11. Συμβαστική Δ πέντε ομάδων που περιλαμβάνει την παραγραφό 4 της, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ψήφι κατά αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Αιτιολογική 12, τροπολογία 2, δεν ψηφίζεται διότι είναι α, γλωσσική. Μετά από το 13 έχουμε τη συμβαστική ε5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το αιτιολογικό 14, F, 5 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά από το 14, συμβαστική G, 5 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά από την αιτιολογική 15, η H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική 16, συμβαστική γιώτα, 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί 236 της ηγητρίας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική 17, 238 της κυρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 εκπίπτει Τελειώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της εκθέσεως και δι ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι, ή μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλες και όλοι, πέρας και εγκρίνεται με 39 λέει πρόεδρος ψήφους υπέρ και 2 κατά. Θα ψηφίσουμε τώρα. Α, υπάρχει ακόμα μια ψηφοφορία. Η τελευταία για το νομοθετικό ψήφισμα. Πρόκειται για νομοθετικό κείμενο. Συμβαίνουν αυτά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Τρίαντα υπέρ, δύο αποχές. Α, όχι, τριάντα πέντε. Ψήφισαν, λέει η πρόεδρος. Τριάντα προς δύο ας βάλουμε μπρος τη μηχανή του χρόνου για να διορθώσουμε, να φτάσουμε στις 36 λοιπόν. Καλά. Τώρα, η απόφαση για την έναρξη των, των ε, διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Η διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελεστεί από την εισηγήτρια, τους σκιώδεις εισηγητές και θα προεδρεύσει η πρόεδρός σας, που σημαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα με τα εξή πρόσωπα. Αγαπητή Μαρία Ναρκίν, Καρή Μαντελή και Γιώργιος Τούσας. Dans le respect des genres. Le mandat Τώρα, το κείμενο θα είναι αυτό που και στο πρώτο τριμερή, ο πρώτος τριμερής διάλογος μάλλον θα γίνει τον Ιανουάριο σε, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί ακόμη σε συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου. Τελειώσαμε τώρα τις ψηφοφορίες και ερχόμαστε στο θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης έκθεση της κυρίας Βερόνικα Λοπέ Φοντανιέ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το 2013. Θα εξετάσουμε φυσικά τις κοινωνικές πτυχές και την απασχόληση. Πρόκειται για έκθεση για την οποία ισχύει ενισχυμένη συνεργασία ή όχι. Όχι, Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, υπάγεται ενισχυμένη συνεργασία και η ΡΕΚΙ θα υποβάλει γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια τις αδερές γραμμές της έκθεσης. Είχαμε ελάχιστο το χρόνο γιατί στις 28 λάβαμε την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και χθε έστειλα το σχέδιο έκθεσης στους συναδέλφους, νομίζω να πρόλαβα να το εκθέτασαν διεξοδικά. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι κοινωνικέ πτυχέ και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γνωρίζοντα, βέβαια ότι η θέση μα δεν αναγνωρίζεται δεόντω δεδομένη τη δημοκρατική νομοποίηση που έχουμε. Χρησιμοποιούμε το τύπο των εκθέσεων ε, ίδιας πρωτοβουλίας ε, δεν πρόκειται για νομοθετική έκθεση, αλλά για κανονική. Συνοδεύεται από παράρτημα με νομοθετικό ψήφισμα και συγκεκριμένες συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ελπίζω να συγκεντρωθεί ευρεία πλειοψηφία και να ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο γνώμη μας. Καταρχήν ξεκινούμε από μια περίπλοκη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που δυστυχώς επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς. Αυξήθηκε η μακροχρόνια ανεργία, αυξήθηκε η ανεργία των νέων και αυξήθηκε ο κοινωνικός αποκλεισμός, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους τομείς και στρώματα της κοινωνίας. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Ε, τα κράτη-μέλη και με τη στρατηγική 2020 και με τις δεσμεύσεις τους δυστυχώς υστερούν σε σχέση με τις συστάσεις που υποβάλαμε για το 2012. Αλλά ούτε τηρήθηκαν οι συστάσεις μας α, της έκθεσης Κορνέλισεν. Γι' αυτό και η δική μου έκθεση που είμαι βέβαια ότι θα εμπλουτιστεί και θα βελτιωθεί χάρη στις δικές σας τροπολογίες απαριθμεί μια σειρά προτεραιοτήτων. Η πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Η εφαρμογή των πολιτικών προσανατολισμών του 2012 στα κράτη-μέλη, γιατί μέχρι στιγμής δεν έληξαν δεόντως υπόψη αυτοί οι προσανατολισμοί, θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η λήψη υπόψη τους για το 2013. Επίσης τα κράτη-μέλη καλό θα ήταν να αναλάβουν τις δεσμεύσεις και να ε, τις περιλάβουν στα προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων για το 2013. Ε, το θέμα της ανεργίας των νέων είναι κέριο και χωρίς κονδύλια πολύ δύσκολα θα καταφέρουν τα κράτη-μέρη να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Δεν ξέρω αν εξαρτάται αυτό από εμά, αλλά στην Επιτροπή Προπολογισμών θα πρέπει να γίνουν τεράστιε προσπάθειε ώστε να εξασφαλιστούν αυτά τα κονδύλια. Δεύτερη προτεραιότητα. Δημιουργία θέσεων εργασία μέσω κάποιων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίαση που θα δημιουργεί πρόσφορο έδαφο για την απασχόληση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα και να θεσπίσουν μέτρα που να δημιουργούν θέσει εργασία και να ενισχύουν τι επιχειρήσει, δημιουργώντα και ε, ε, πρόσβαση των, μικροεπιχειρήσεων, ε, των επιχει... μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και δημιουργώντας πρόσφορο κλίμα και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Μιλήσαμε επίσης για τις φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις απασχόλησης ε, που είναι πολύ ποιοτικέ. Άλλο θέμα, σημαντική προτεραιότητα, η ανεργία των νέων, μεγάλη μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα στην Ισπανία είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τα προγράμματα μαθητείας, κατάρτισης, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των νέων στην παιδεία και στην επαγγελματική επιμόρφωση και να δοθούν ε, ενάψματα σε επιχειρήσεις για να συμπεριλάβουν νέους ε, στα προγράμματα αυτά και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες στρατηγικές για, την, για τους άνεργους νέους στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για τους ανειδίκευτους. Επίσης, χρειάζονται κονδύλια για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Τέταρτη σημαντική προτεραιότητα. Αγορές ε, πιο ευπροσάρμοστες, δυναμικές, ε, ε, που δεν θα αποκλείουν κανέναν και θα εξασφαλίσουν ποιοτικέ θέσει απασχόλησης. Να προβλέψουμε προϋποθέσεις ώστε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών, των αναπήρων και των ανθρώπων που χρειάζονται που είναι πιο ευάλωτοι και χρειάζονται οπωσδήποτε μία θέση εργασία κάτι που δεν ελήφθη όντως υπόψη μέχρι στιγμή. Οι αγορέ εργασία θα πρέπει να είναι πιο προσάρμοστες, πιο δυναμικέ και να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ των μέτρων λιτότητα που είναι απαραίτητα, αλλά που δεν θα πρέπει να αποβαίνουν ει βάρο τη ποιότητα ε, τη απασχόλησης και τη ε, προστασία ε, των εργαζομένων και των κοινωνικών του δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και το σημείο αυτό πέμπτη προτεραιότητα. Κοινωνική ένδυα και κοινωνικός αποκλεισμός. Πρέπει να επαγρυπνούμε και παρά την έμφαση που δίνει το σημείο αυτό να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτο σημείο. Δημοκρατική νομιμοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Το δηλώσαμε επανειλημμένο. Αν θέλουμε οι συμπολίτε μα να πιστέψουν στι μεταρρυθμίσει και στα μέτρα παρόλο που θα είναι μέτρα λιτότητας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και τέλος, θα πρέπει με αναλογικό και διαφοροποιημένο τρόπο να αναζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους ε, για τη δημοσιονομική εξυγίαση με τρόπο που θα εξασφαλίζει και την ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Να μην επιμένουμε μόνο στα μέτρα λιτότητας. Είναι ένα απαραίτητα, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται εις βάρος της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. Προσπάθησα εν συντομία να παρουσιάσω τις αδρές γραμμές της έκθεσης που είναι αρκετά διεξοδική. Φυσικά θα τροποποιηθεί με τις τροπολογίες. Είχαμε ελάχιστο χρόνο για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης. Ελάχιστο χρόνο έχουμε και για τις τροπολογίες δυστυχώς, αλλά πιστεύω ότι χάρη σε αυτές θα εμπλουτιστεί και θα βελτιωθεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σέρτζο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την κυρία Λόπε Φοντάνια για την αξιόλογη έκθεσή της. Η ομάδα μας είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την εισηγήτρια προκειμένου να καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, διεκδικήσεις και έμφαση σε ορισμένα σημεία. Το σχέδιο έκθεση είναι πολύ καλό σημείο αφετηρία. Και δεν μας δημιουργεί τόσο πρόβλημα η έκθεση, όσο η ανακοίνωση Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Βέβαια δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερα μετά την παρέμβαση του Όλη Ρέν της περασμένης εβδομάδας. Γιατί δυστυχώ δεν αλλάζει η πορεία που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μία ακόμη χρονιά που βυθιζόμαστε όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική η πολιτική της. Γιατί αυτό χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτε να αποδείξουμε ότι οι πολιτικές μας είναι αποτελεσματικές. Έχουμε όμω την τρίτη ετήσια επισκόπηση για τη ανάπτυξη, την τρίτη αυτή έρευνα και μελέτη και διαρωτόμαστε πού βρίσκεται, πού είναι σήμερα η ανάπτυξη. Γιατί δεν βλέπουμε καμία τόνωση ανάπτυξη. Τέσσερα χρόνια προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κρίση, να κάνουμε διεξοδικές αναλύσεις, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την τρίτη ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης παρουσιάζει τρεις στόχους. Διατείνεται ότι ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα. Πώς όμως, γιατί αν η μόνη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα είναι η μείωση του μισθολογικού κόστου των επιχειρήσεων και η μείωση κατά 20% των μισθών στις χώρες, κατά μέσο όρο, αν βγάλει στο δρόμο του ε, τους εργαζόμενους ή καταργήσει τις συλλογικέ συμβάσεις, ελαστικοποιώντα ελαστικοποιώντας την αγορά, ναι μεν θα κερδίσουμε σε ανταγωνιστικότητα, αλλά θα καταβαραθρώσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Και αν δώσουμε περισσότερη έμφαση στα ε, μισθοδοτικά μοντέλα και όχι στο παραγωγικό μοντέλο, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από την κρίση. Και σίγουρα δεν θέλουμε την ανταγωνιστικότητα πάση θυσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι μειώθηκαν οι εντάσεις στο χρηματοπιστωτικό κόσμο. Πολύ υποπτό μου φαίνεται αυτό. Γιατί όταν ακόμη και σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καμία πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Έχουμε τρεις χώρες ε, ε, που έχουν τεράστια spread, γύρω στα 400, 400 μονάδες σε σχέση με το γερμανικό επιτόκιο, που βρίσκονται στα πρόθυρα της διάσωσης και πολύ αρνητικές προοπτικές για την ανάπτυξη. Πού είναι αυτή η μείωση των ε, εντάσεων και των τριβών χρηματοπιστωτικές αγορές που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφωνούμε ως προς αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια τριετή εφαρμογή εσφαλμένης στρατηγικής Φυσικά δεν μιλάει για επιτυχία στην ε, ε, απασχόληση, γιατί δεν υπάρχει, ούτε για τη μείωση της φτώχειας, είτε το αποκλεισμό αλλά μιλάει για τη μείωση των εμπορικών ελλημάτων κάποιων χωρών. Αλλά και αυτό παγίδα είναι. Μειώνονται βέβαια τα εμπορικά ελλείμματα, γιατί αυξάνονται κάπως οι εξαγωγές, αλλά τι γίνεται με την παραγωγή. Στις 20 σελίδες της ετήσιας επισκόπης ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε μια φορά δεν κάνει λόγο για το τι μπορούν να κάνουν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουν το εσωτερικό εμπόριο, την εσωτερική ζήτηση και να αυξηθεί το μισθολογικό κόστος. Γιατί αν η Γερμανία αυξήσει κατά 5-10% του πάγιου μισθολογικού κόστους, θα βελτιωνόταν η κατάσταση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχυόταν η ανάπτυξη. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για κοινή ευθύνη, αλλά είναι άνηση η κατανομή αυτή τη ευθύνη. Και μεταξύ των χωρών μελών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι χώρες τηρούν τις συστάσεις που τους γίνονται, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις τους οδηγούν σε κοινωνική ασφυξία. Αλλά τι γίνεται με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Πού είναι εκεί το αναπτυξιακό σχέδιο που μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Τραπεζική Ένωση, τα ευρωμόλογα, τα επενδυτικά έργα. Είναι κοινή, επιμερισμένη ευθύνη. Και οι δεσμεύσει θα πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η στρατηγική λιτότητα καταπνίγει την ανάπτυξη και ενισχύει την ανεργία και τη φτώχεια. Τα αναγνωρίζει μεν αυτά και αναγνωρίζει ουσιαστικά την αποτυχία της πολιτικής της, αλλά ταυτόχρονα δεν αλλάζει άρδιν την πολιτική αυτή και τη συνεχίζει με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμη και μεγαλύτερη ανεργία και φτώχεια. Επίσης μιλάει για δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές που θεωρεί ότι είναι αποκλίνοντες. Θεωρεί όμως ότι η μείωση της δαπάνης είναι σημαντικότερη από την αύξηση των εσόδων. Ναι με να προσπαθήσουμε να περικόψουμε κάποιες δαπάνες, αλλά γίνεται άνηση περικοπή στα κρατη και δεν αναφέρεται ιδιαίτερα η παιδεία, οι παραγωγικές επενδύσεις, η υγεία, γιατί δεν είναι όλες οι δαπάνες ίδιες, ούτε θα πρέπει να περικόπτονται με τον ίδιο τρόπο. Και μπορούμε να έχουμε μια αύξηση των εσόδων, όχι όμως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πλουσίων. Θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση εδώ και διακρίσεις, γιατί είναι πολύ γενικές αυτές οι παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γιατί αυτή η ιδεολειψία με τον οδικό χάρτη για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Είναι σαν ταινία τρόμου αυτό το δημόσιο έλλειμμα. Να το μειώσουμε μεν, αλλά προσοχή στο χρονοδιάγραμμα. Αλλά όπως γίνεται και με τις δίαιτες, όταν κανείς θέλει να δυνατήσει, θα πρέπει να το κάνει σταδιακά. Δεν μπορεί μέσα σε τρεις μήνες να χάσει 50 κιλά διακυβεύει την ίδια του την υγεία και την απειλή. Προσοχή λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τη μείωση του ελλείμματο. Μα λένε οι οικονομολόγοι, αν, αν επιμηκύνουμε το χρονοδιάγραμμα μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματο, τηρώντα το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη και τηρώντα και το εξαπλό πακέτο, θα μπορούσαμε κάθε χρόνο να εξοικονομούμε 800 δισεκατομμύρια Ε, γιατί λοιπόν αυτή η ιδεολειψία ε, και η ακαμψία να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω ε, ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε και το χρυσό κανόνα που το αναφέρει και η Βερόνικα στην έκθεσή της και να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων επενδύσεων. Μερικές επενδύσεις όπως αυτές στην υγεία και την παιδεία δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επίσης, έχουμε πολλά στοιχεία στο κεφάλαιο απασχόληση. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε στην Επιτροπή μας και τα έχουμε όχι μόνο στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη, αλλά και στις δικές μας εκθέσεις. Ωραίες υποσχέσεις, τις κάνουμε κάθε χρόνο, τις ανανεώνουμε, αλλά δεν τηρούνται. Ούτε κανένας αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την τήρησή τους. γιατί φαίνεται ότι είναι καλοπιστικές μερικές φορές ε, οι προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην Επιτροπή Απασχόλησης χρόνια ολόκληρα λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα εθνικά προγράμματα απασχόλησης. Αλλά δεν γίνεται καμία ε, επιτήρηση. Δεν ξέρουμε τι προγράμματα εφαρμόζονται κάθε χρόνο. Ποιοι είναι οι στόχοι του. Μόνο το συνολικό ποσό γνωρίζουμε. Που είναι εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Φέτος στην Ισπανία μειώθηκε το 60% του προϋπολογισμού τους και κανένας δεν είπε τίποτα. Από 8 δισεκατομμύρια μειώθηκε ο προπολογισμό σε 3 δις και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Τι γίνεται με τη διαβίου κατάρτιση, την επαγγελματική επιμόρφωση ή την αναδιάρθρωση του Ταμείου Συνοχής. Πώς θα μπορέσουμε με όλα αυτά τα μέτρα να ενισχύσουμε την απασχόληση και ιδιαίτερα στους νέους που μαστίζονται από την ανεργία. Δεν μπορούμε να δίνουμε έναν Άγιο για να αντίσουμε άλλον. Το Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο καλό θα είναι να είναι απαιτητικά στους στόχους τους και να ελέγχουν την αξιοποίηση των κονδύλιων, αλλά χρειαζόμαστε και νέα κονδύλια, γιατί έχουμε ένα ιστορική σημασία πρόγραμμα για την απασχόληση, σε μια κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή δεν μπορούμε να αρκεστούμε στους μηχανισμούς και στα κονδύλια που είχαμε μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς και νέα κονδύλια και να είμαστε και πιο απαιτητικοί οι ίδιοι με τους εαυτούς μας. Και κάποιες σοβαρές ανησυχίες. Με ανησυχεί η έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αγορές εργασίας. Τις θεωρεί τη μοναδική ε, σχεδόν διέξοδο από την κρίση. Και με ανησυχούν κάποιες φράσεις όπως ότι είναι απαραίτητο να μειώσουμε τις αποζημιώσεις στις στερεότυπες συμβάσεις. Η αποζημίωση λόγω απόλυση δεν έχει σχέση με την απασχόληση. Και με ανησυχεί αυτό που το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, μιλάμε για τις στερεότυπες συμβάσεις. Ε, αναλύθηκαν ε, διεξοδικά οι άτυπικές συμβάσεις, άτυπες συμβάσεις τι έγινε με την κρατικοποίηση των τραπεζών. Εκεί είχαμε μισθολογικές, ε, εργασιακές μάλλον μεταρρυθμίσεις που στέρισαν από τους εργαζομένους τα μισά τους δικαιώματα, ιδιαίτερα στις αποζημιώσεις για, για Τι έγινε με τις τράπεζες. Κρατικοποίησαμε μερικές τράπεζες και μάλιστα με κοινοτικά κονδύλια. Αλλά ουσιαστικά απολύονται οι εργαζόμενοι χωρίς καμία αποζημίωση. Ενώ τα διοικητικά στελέχη λαμβάνουν παχυλές αποζημιώσεις με σκανδαλώδεις αποδοχές αστρονομικές, ενώ μαζικά απολύονται από τις κρατικοποιημένες αυτές τράπεζες χωρίς κανένα δικαίωμα οι εργαζόμενοι τους. Τι γίνεται με τις ρήτρες συλλογικών συμβάσεων. Δεν μπορούμε να τις αποδυναμώνουμε συνέχεια. Με ανησυχεί και η απέτηση της μείωσης του φορολογικού βάρους, ιδιαίτερα λόγω της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε να μειώνουμε το, το δημοσιονομικό έλλειμμα εις βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, ε, για τις εγγύησεις των νέων, να μην ξεχνούμε την ποιότητα στην απασχόληση, γιατί χωρίς ποιοτικέ θέσει εργασία θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Κυρία Λόπε Φοντανιέ, πολύ καλή αφετηρία βέβαια, αλλά η η στρατηγική αυτή μου φαίνεται ως ε, ωραία λόγια, πεπτερώνεται και βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά ελάχιστα από τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Μάριαν Χάρκιν και μετά Κορνέλισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δύο συνάδελφοι τα είπαν όλα. Δεν έμεινε και τίποτα να πολύ να πω. Ωστόσο, θα κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Δυστυχώ, μόλι σήμερα το πρωί την είδα, οπότε ε, έριξα μια γρήγορη ματιά, αλλά φαίνεται να τα περιλαμβάνει όλα και όπως και οι συνάδελφοι θα ήθελα να το μελετήσω περισσότερο. Συμφωνώ με τα μηνύματα αυτά. Πιστεύω πως είναι στεναρά και ίσω όντω και να πρέπει να ενισχυθεί κάπω η παράγραφο 3. Και πάλι Μιλάτε για το γεγονός ότι αυτοί οι στόχοι σημερινοί δεν ε, πετυχάνονται και για το 2020 και για την προσθέμενη αξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όντως θα πρέπει να ε, παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη συνολικά προγράμματα, εθνικά προγράμματα και είναι απογοητευτικό το ότι δεν έχει συμβεί. Εδώ βλέπουμε βέβαια τη γενική εικόνα και όχι την εθνική. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συζήτηση με τους επιτρέπους Ρεν και Άντορ για την ετήσια ε, έρευνα για την ανάπτυξη και θα πρέπει να σας πω ότι δεν ε, έμεινα πολύ ικανοποιημένη γιατί δεν έχουμε αποδείξεις για το ότι λειτουργεί η πολιτική. Λειτουργεί σε κάποιους ε, τομείς και όχι σε άλλους. Και αν δούμε την πολιτική λιτότητα. τι γίνεται, τελικά τα ελλείμματα έχουν <coughs> συγγνώμη, τα χρέη έχουν αυξηθεί περισσότερο από όταν ξεκίνησαν οι πολιτικές αυτές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη αυτά να ε, καλύψουν τα χρέη και να μειώσουν τα επίπεδα ε, αντίστοιχα με την ανάπτυξή τους. Πιστεύω πως η Κομισιόν και με τη στήριξη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να δει με φρέσκια ορμή το τι κάνουν. Δεν λέω να αλλάξουν εντελώ πορεία 180 μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως λιγότερο τα χρονοδιαγράμματα, να, βγούμε, να βγάλουμε τις παροπίδες, να μην είμαστε προσιλωμένοι αυστηρά σε, μια, σε ένα στόχο. Ξέρω ότι δεν μιλάει μόνο για λιτότητα, δεν θέλω να είμαι άδικη προς την Κομισιόν, αλλά ο πυρήνα είναι βασικά λιτότητα Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές που θα δώσουν στα κράτη-μέλη που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση μια ευκαιρία να βγουν από αυτή την κατάσταση. Χτες για παράδειγμα, και είμαι βέβαιη πως αρκετοί θα ήσασταν εκεί, πήγα στην διάσκεψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πραγματικά ήταν σπαραξικάρδιο να ακούμε τι είχαν να πούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο από τα κράτη-μέλη που ε, αυτή τη στιγμή έχουν βάλει τον κορσέ τη αλλά και από άλλα κράτη-μέλη όπου πραγματικά έχουν χάσει τελείως τις δυνατότητές τους, να έχουν ανεξάρτητη σία από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουν αξιοπρέπεια και αυτό είναι ο των πολιτικών που εμεί. Ε, συνεχίζουμε. Θα πρέπει να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά, να τα αντισταθμίσουμε κάπως. Ιδιαίτερα στις παραγράφους 25-26 που λέτε πως ναι, μεν πρέπει να γίνει εξυγίαση, να συνεχιστεί, αλλά σε με αναλογικό και πιο φιλικό τρόπο. Αν μπορούσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό θα ήταν χρήσιμο και ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και στα κρατημέλη και να ολοκληρώσω λέγοντας πως συμφωνώ με το τελευταίο τμήμα που μιλάτε για αυξημένο δημοκρατικό έλεγχο, εποπτεία και ε, ιδιοποίηση όλων αυτών γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα κρατημέλη αλλά ιδιαίτερα σε καποια κρατημέλη οι πολίτες αποξενώνονται από την Ενένωση και από το τι κάνει, γιατί το μόνο που βλέπουν είναι οι τίτλοι των εφημερίδων. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν το Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν να παίξουν ένα πιο σημαντικό ρόλο, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται πιο πολύ σύνδεση με την Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι. Merci Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κορνέλισεν και μετά η κυρία Ζούμπερα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας ε, την ε, εισηγήτρια που έφτιαξε ε, τόσο περιεκτικό σχέδιο έκθεσης σε τόσο σύντομο χρονικά διάστημα. Ξέρω πόσο σκληρή δουλειά ήταν την περασμένη φορά να τα καταφέρουμε στην ώρα που έπρεπε και πιστεύω τα πήγατε πολύ καλά. Είναι μια ευκαιρία να έχουμε μια πραγματικά γενική συζήτηση για τη... το τι θα πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από την κρίση. Με λύπησε που πέρυσι για την έκθεση, την αιτήσια για την ανάπτυξη ή το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, δεν ελήφθησαν πολλά υπόψη. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητο η δημοκρατική νομιμότητα να χαράζουν την κατεύθυνση που θα πάρουν οι οικονομίες τους. Ε, δεν μετράει και τόσο πολύ και νομίζω πως κάνουν λάθος. Είμαι ευτυχής για τη μορφή που διαλέξατε για αυτή την έκθεση, είναι διαφορετική. Στην ουσία αναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να τη δράσει στα όσα λέμε αυτή τη φορά. Γιατί από μόνοι τους δεν δείχνουν προθυμία να δεχτούν ε, τα όσα τους προτείνουμε. Είμαι ευτυχής γιατί αναφέρονται οι προτεραιότητε για το 2020 και ότι δεν φτάνουμε κοντά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αντίθετα, απομακρυνόμαστε. Η ανεργία έχει αυξηθεί, η ευτόχεια έχει αυξηθεί, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια παραπάνω φτωχοί. Περικοπές του προπολογισμού γίνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ αυτός υποτίθεται θα ήταν ένας τομέας ε, που θα γίνονταν επενδύσεις ώστε να προωθηθεί καινοτόμα οικονομία. Πυροβελοντικοί στόχοι παραβλέπονται, παραμελώνται και δεν φτιάχνονται νέε θέσεις πράσινης απασχόλησης. Μας περιπτώσει το 2000, η ατζέντα του 2020 φαίνεται να έχει βγει από τους τίτλους πλέον και από τις προτεραιότητες. Δηλαδή ποια είναι η φιλοσοφία, ότι όλα καλά από τη στιγμή που έχουμε λεφτά και η οικονομία πάει καλά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή, τα έχουμε όλα αναστείλει μέχρι ότου να βγούμε από την κρίση. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από την κρίση αν δεν αρχίσουμε να φτιάχνουμε πάλι θέσεις εργασίας στον πράσινο τομέα. Και θα ήθελα Να σας πω ότι εκείνο το κομμάτι για την κοινοβουλευτική συμμετοχή και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ισχυρό. Αυτά. Σας ευχαριστώ. κυρία Ζούμπερ. Και μετά δύο λόγια που θα πω κι εγώ πριν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Όχι. Λοιπόν, κλείνω το λόγο των ομιλητών. Η κυρία Ζούμπερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω το έγγραφο το οποίο επεξεργαστήκατε γιατί έφτασε χθε το βράδυ. Αλλά πρόσεξα πολύ την παρέμβασή σας, την εισήγησή σας και αναφέρατε και θέλω να προσπαθήσω να καταλάβω πώς γίνεται αυτή η έκφραση συγκεκριμενοποιείται στην πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά δυσκολεύομαι να την κατανοήσω. Και αυτό που είπατε ήταν να διατηρηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση με στόχο την ανάπτυξη. Γιατί αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ότι η η δημοσιονομική εξυγίανση μετατρέπεται σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Και σκεφτόμουν λοιπόν τη χώρα μου, όπου οι πολιτικές εξυγίανσης εφαρμόζονται μεταφράζονται σε ένα ε, ε, πολύ σκληρό πρόγραμμα λιτότητας ε, από την Τρόικα αλλά στην επασχόληση τι έγινε. Μείωση του κόστους ε, της μονάδας ε, εργασίας και ε, λιτότητα, τρομερή λιτότητα. Επίσης καταργήθηκαν τα διάφορα επιδόματα των διακοπών και τα λοιπά και απολύθηκε πολλοί κόσμος και στη δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, για τον επόμενο χρόνο θα απολυθούν το 50% των συμβασιούχων του δημόσιου τομέα, που σημαίνει τη μεγαλύτερη μαζική απόλυση ανθρώπων που έχει γίνει ποτέ. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική εξυγίανση. Και χτες άκουγα τα νέα και μάλιστα άκουσα ότι από αυτό το Σεπτέμβριο, το φετινό Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα στην Πορτογαλία, οι πωλήσει ε, στην λιανική πώληση μειώθηκαν κατά 4,5%. Το περισσότερο ποσοστό δηλαδή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, άρα λοιπόν κάνει οικονομία, πάβει να αγοράζει και εφόσον δεν αγοράζει καταστρέφονται και διαλύονται καθημερινά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ειλικρινά η δυσκολία μου είναι να καταλάβω Πώς γίνεται να συνδυαστούν τα δυο αυτά. Γιατί εντάξει τα λόγια είναι λόγια, αλλά στην πράξη ε, όλα αυτά έχουν συνέπειες. Θα υποβάλουμε τροπολογίες, εγώ θα υποβάλω τροπολογίες και μία από τις προτάσεις που θα κάνω θα είναι ακριβώς μια πρόταση αντίθετη που αναφέρεται στο θέμα του στόχου αξιοποίησης των, των μισθών, δηλαδή μάλλον ε, των μισθών. Όχι ως μορφή κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά ως μορφή ενδυνάμωσης της οικονομίας μας. Και ελπίζω ότι θα δεχτείτε τις προτάσεις που θα σας υποβάλω. Ευχαριστώ. Euh, euh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να πω ότι πιστεύω πως το σύνολο των συναδέλφων που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα το γνωρίζουν. Να πούμε δηλαδή πόσο αυτό αυτή η όλη υπόθεση είναι σημαντική και η Κομισιόν καλά θα κάνει να λάβει υπόψη, μάλλον σοφά ε, δέχτηκε την ε, άποψή μας που αλλάζει τον τίτλο ήδη της πρότασης, γιατί όταν ε, μας προτείνεται μια ετήσια ξέταση της ανάπτυξης, ε, είναι κάπως παράδοξο να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τις αναλύσεις ε, που έχουν γίνει από διάφορους ε, και από την ομάδα στην οποία ανήκω. Ε, καλό λοιπόν όλους να δείτε αυτό το έγγραφο, να το διαβάσετε. Η σοσιαλιστική ομάδα όπως θα το έχετε διαπιστώσει, έχει αναθέσει σε τρεις ανεξάρτητες σε τρία ανεξάρτητα Ινστιτούτα να κάνουν ε, μελέτη της ανάπτυξης. Και τελικά, δηλαδή να κάνουν μια αποτύπωση τη της Γιατί μια από τις δυσκολίες τη συζήτηση που έχουμε και που αυτή τη στιγμή και που επιδεινώνεται με τις, ε, μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου της επόμενης εβδομάδας σήμερα, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και επί τη ουσία. βλέπουμε μόνο μία στρατηγική να έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή, ο φεντεραλισμός περιορίζεται ε, σε ανταλλαγές απόψεων μεταξύ Κομισιών και ΔΕΚ και Κομισιών. Όμως η συζήτηση ανάμεσα στο Εθνικά Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό δεν, θα, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο ο φεντεραλισμός μόνο με τον κανόνα της πειθαρχία, της ποινή, της κύρωσης και της λιτότητας. Έπειτα, βλέπουμε αυτή την εικόνα της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη. Υπάρχουν οι προτάσεις της Κομισιόν για να φτιαχτεί αυτό το περίφημο ε, συμβόλαιο από πάνω δηλαδή θα ερχόταν. Έχουμε δηλαδή τις συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα, έχουμε το αναρτήσιο δικό χάρτη και όλα αυτά από πάνω μέσα σε, μια, σε ένα συμβόλαιο που επίσης θα είναι συμβόλαιο ε, τιμωρίας στην ουσία κυρωτικό. Ε, εντάξει, τα, κάποια κράτη-μέλη παραστράτησαν, ε, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε κτλ. Αλλά δεν νομίζω πως το φάρμακο είναι καλύτερο από το, τα λάθη που έκαναν. Υπάρχουν εδώ και δύο διαστάσεις οι οποίες καθόλου δεν αναφέρονται εδώ που είναι η κοινωνική και αν δούμε στην ετήσια εξέταση της ανάπτυξης, ναι βεβαίως ε, πιστεύω ότι για την ε, Επιτροπή μας, για τα όσα είδαμε, για την απασχόληση των νέων, για το γεγονός υπάρχει ιδέα ότι στις ε, επενδύσεις στο εθνικό και στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι μεγάλη Ε, η συμμετοχή είναι ένα επιχείρημα αυτό το οποίο θα πρέπει να, στηρίξουμε και η έκθεσή σας ε, θα πρέπει να μας βοηθήσει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και να προχωρήσουμε και πιο πέρα γιατί Η Γενική Διεύθυνση ΦΙΝ είναι πραγματικά ε, εξαιρετικά μεγάλη και ανάμεσα στην ΕΠΣΚΟ και στο ΕΚΟΦΗΝ βλέπουμε και στο Συμβούλιο πως η ισορροπία είναι ανύπαρκτη. Και Το θέμα της ισορροπίας πρέπει να αφορά και την ανομοιογένεια των χωρών. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την ε, σφαιρική κατάσταση, αλλά μετά ανακράτως μέλος πρέπει να δούμε τι τρέχει. Και δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τα ίδια πράγματα σε όλους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μακροοικονομικές ε, διαφορές που πρέπει να καταπολεμήσουμε και να διορθώσουμε. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν έχω την εντύπωση ότι είναι σε μια σε μια έτσι μονομερή προσέγγιση. Ε, μιλάμε για ηθικό κίνδυνο. Κανένας δεν μιλάει βέβαια για ποινή, για τιμωρία. Αυτά ήθελα να πω. Και η Κομισιόν εδώ αντιπροσωπεύεται από τον κύριο Λορέν Γκαρσία και η τον κύριο Άγκστετ. Ποιος από τους δύο θέλει να πάρει το λόγο. Αλλά έχει το λόγο η Κομισιόν. Καλημέρα σας, Σαντιάχο Λοράνκα. DG Employment, απασχόληση. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να πω δύο λόγια στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Σίγουρα το γενικότερο πλαίσιο δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Είδαμε πως ε, έχει υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω πως όλα αυτά αντιπροσωπεύονται αρκετά καλά στην ε, συζήτηση και στην ετήσια έκθεση περί ανάπτυξης η κατάσταση είναι δύσκολη και είναι και διαφορετική, διαφοροποιημένη. Επιδεινώνεται εν γέννη, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία καταστάσεων που αντικατοπτρίζεται και στα διαφορετικά ποσοστά ανάπτυξης, όπου ορισμένε φορές είναι ψηλότερη η αρνητική ανάπτυξη. Και έχουμε και πολύ διαφορετική κατάσταση στην αγορά εργασίας και αυτό είναι πολύ ορατό όσον αφορά τα διάφορα ποσοστά ανεργίας. Και αυτό το βλέπουμε και στην έκθεση. Αυτή η διαφορά της κατάστασης στις αγορές εργασίας αντικατοπτρίζεται και σε κάτι που αναφέρθηκε σε διάφορες ευκαιρίες σήμερα και αφορά την εξυγίανση της οικονομίας και το πιθανό περιθώριο ελιγμό για τα διάφορα σε μια κατάσταση όπου ή διαφορετι... διαφοροποίηση αφορά δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, περιθώριο λιγμού και δεύτερον, την ανάγκες μόχλευσης της οικονομίας που αντικατοπτρίζονται είτε από τη δημόσια χρέωση είτε από την ιδιωτική χρέωση. Αυτά τα εξετάζουμε για ταυτόχρονα με τις ανάγκες αποκατάστασης της δυνατότητας δανεισμού της οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε διαφοροποιημένους δρόμους για την εξυγίανση και υπάρχει και διαφορετικός χώρος περιθώριο λιγμού ανάλογα με το κράτος μέλος και αυτό ήδη αντικατοπτρίζεται σε κάποιες αποφάσεις που ε, <clears throat> έχουν ληφθεί ότι δηλαδή πρέπει να διαφοροποιηθεί η προσέγγιση. Είδαμε και γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη να διατηρηθούν διάφορα στοιχεία κατά την εφαρμογή της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η Κομισιόν ήταν σαφής στον εντοπισμό διάφορων θεμάτων για την ε, πολιτική και πρέπει όντως να ενισχύσουμε την αποκάλυψη και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και σίγουρα θα πρέπει να φροντίσουμε για την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συστημάτων που είναι ύψης της σημασίας ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Γνωρίζουμε όμως τις ανάγκες, γνωρίζουμε το ε, τμήμα απασχόλησης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης που ήταν ε, το αντίστοιχο του εθνικού σχεδίου για φέτο και προγραμματίζουμε να στείλουμε πιο λεπτομέρη καθοδήγηση στα κρατημέλη για την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης ώστε να περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το τι θα, θα περιλαμβάνεται στα εθνικά προγράμματα για ε, τον... τις θέσεις απασχόλησης. Εν τω μεταξύ, κάποιε από τι προτεραιότητε κλειδιά έχουν ε, βαθεθεί περισσότερο από πλευρά κομισιών με βάση το πρόγραμμα ε, εγγύηση των νέων για την απασχόληση των νέων. Και υπάρχει μια λεπτή ισορροπία φυσικά όσον αφορά την ανάγκη προστασίας διατήρησης των κοινωνικών συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και της ανάγκης των ε, μειονεκτικών ομάδων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγένσης. Θα σταθώ σε αυτά και φυσικά θα είμαστε ε, θα συνεργαστούμε με τον εισηγήτρια και τις ομάδες αν χρειάζονται διευκρινήσεις για οποιαδήποτε πτυχή της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ η εισηγήτρια. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους και οδησηγητές αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προθυμία που εξέφρασε για διάλογο μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα απαντήσω τώρα. Προτιμώ να αφήσω χρόνο στους συναδέλφους να μελετήσουν ε, προσεκτικά την έκθεση και νομίζω ότι είναι απολύτω απαραίτητο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γιατί αν θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας, χρειαζόμαστε ευρεία πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. <laughs> Θέλουμε ένα κείμενο που θα το υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική δυνατόν πλειοψηφία. Έτσι θα δώσουμε ένα χειρό μήνυμα και θα ακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών. Βραχύτατη. Όπως ήταν και για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης. 13 Δεκεμβρίου το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 18 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 14 Ιανουαρίου. Στο Στρασβούργο. Ενώ στις 4 και 5 Φεβρουαρίου θα εξεταστεί και θα ψηφιστεί η έκθεση στην Ολομέλεια. Στις 28 Ιανουαρίου θα έχουμε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Πολύ σημαντικό ραντεβού για τη διαπραγματευτική μας ομάδα. Γιατί εκεί θα έχουμε μια συνεννόηση για τα θέματα αυτά με τους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης. Το σημείο 11. au point 12, pardon. Euh, Όχι, το 11 το κάναμε. 12, 12 εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαία και την εφαρμογή της οδηγίας 2009-13 για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΞΑ, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές, σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και τροποποίηση της οδηγίας 1999-63. Έχω λάβει για το σχέδιο έκθεση αυτό οκτώ τροπολογίες. Θα τις σχολιάσω εντός ολίγου. Όπως είπαμε, κατά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, η βασική δυσκολία μας εδώ έγκυται όχι στην ερμηνεία της ε, συνθήκης για την αυτική εργασία, αλλά στους ε, όρους εφαρμογής της στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, δεδομένων των αρμοδιοτήτων αφενός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου των κρατών μελών. Πολλό δε μάλλον που από νομική άποψη μία από τις βασικές καινοτομίες ε, της Σύμβασης για την Αυτική Εργασία προβλέπει ότι άσχετα με την πορεία κύρωσης αυτής της σύμβασης, εφόσον γίνεται επιθεώρηση έλεγχος ένα σκάφος, το κράτος ε, του λιμανιού μπορεί να δεξαγάγει ελέγχους άσχετα από το αν έχει ε, το κράτος σημαίας κυρώσει ή όχι τη σύμβαση από την άποψη διενέργειας ελέγχων διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ χρήσιμη μια τέτοια σύμβαση. Όμως προσκρούμε στο γεγονός ότι η οργάνωση των ελέγχων δεν εμπίπτει σε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στις εθνικές αρμοδιότητες. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια και για τον έλεγχο, αλλά και για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που θα πρέπει να συνοδεύει αυτούς τους ελέγχους. Το σημείο αυτό εξετάστηκε στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη είναι πολύ αποφασιστικά να εμείνουν στις θέσεις τους και αποφασισμένα. Ε, Φιλίπ Τεμπακέρ, Φιλίπ Μπενιόν και Κεζίν Μεσνέρ έχουν υποβάλει τροπολογίες τις 64, 65, 66, 67 που αφορούν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, την κινητοποίηση των κρατών μελών για την ε, άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό Εφόσον οι τροπολογίες αυτές μας βγάλουν από την αντίφαση και το διέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε, θα τις δεχτώ. Αν δηλαδή καταφέρουμε με τις τροπολογίες να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση απέναντι στο Συμβούλιο και να λύσουμε το πρόβλημα, θα τις δεχτώ πολύ ευχαρίστως. Υπό τον όμως ότι θα υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Αλλιώς θα πρέπει να δούμε τι άλλες εναλλακτικέ λύσεις έχουμε για να μείνουμε σταθεροί απέναντι στο Συμβούλιο και να υπερβούμε και το νομικό κόλλημα που αντιμετωπίζουμε. Μία τροπολογία προβλέπει ε, διάλειμμα, μία προθεσμία μεταξύ των ελέγχων, μία ελάχιστη προθεσμία χρήσιμη αυτή η πρόταση γιατί προς το παρόν δεν προσδιορίζεται κάτι στο κείμενο. Αυτό προβλέπει η τροπολογία 66. Τώρα, οι τροπολογίε τη Αγίπτα Στάινρικ διέπονται από την ίδια ιδέα ουσιαστικά. Δηλαδή το θέμα της κινητοποίησης των κρατών μελών για την άσκηση των ευθυνών τους. Χρήσιμες λοιπόν και οι τροπολογίες της κυρίας Στάινρουκ. Βέβαια η τροπολογία 71 που προβλέπει μια ρήτρα ε, είναι σημαντική γιατί θα πρέπει να έχουμε περισσότερη επιρροή στο θέμα εφαρμογής της σύμβασης αυτής από τα κράτη-μέλη. Αυτά. Ελπίζω να σας κατατόπισα. και περιμένω τις παρατηρήσεις σας για τα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης των τροπολογιών. Φιλιππινιό. Um, Έχω μια δήλωση του Φίλντε Μπάκερ που είναι ο σκιώδης ηγητής και δεν έχει προφτάσει να έρθει ακόμη. Απλώς λοιπόν θα διαβάσω τι έχει γράψει. Πρώτα, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεση. Δεν υπάρχουν τροπολογίες πολλές. Μαζί με τον κύριο Μπένιον, δηλαδή εμένα, έχουμε υποβάλει ορισμένε τροπολογίες. Θεωρούμε ότι η Κομισιόν έχει καταθέσει μια καλή πρόταση. Υποθέτω ότι έχουν κάνει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη πριν καταθέσουν τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να δεχτούμε την ε, Οδηγία 2009-13 και την συμφωνία που εφαρμόζει. Δεν θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν ε, τμήματα της Maritime Convention για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να γίνει δεχτή αυτή η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων υποστηρίζοντας επομένω την ε, πρόταση τη Κομισιόν και προσθέτοντα όσο δυνατόν λιγότερα. Έχω ορισμένε τροπολογίε για την πιστοποίηση που ε, λαμβάνουν υπόψη και ορισμένε τροπολογίε του εισηγητού για να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με την πρόταση τη Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομική βάση για να επιβάλλει απαιτήσει πιστοποίηση. Αυτά ε, διαλαμβάνονται μόνο στην διεθνή ναυτική νομοθεσία. Η πρόταση της Κομισιόν στοχεύει στην επιβολή της συμφωνίας των ε, εταίρων. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομική βάση για την έκδοση πιστοποιητικών και ιδίως ναυτικών. Ήδη στην οδηγία 2009-13 περιλαμβάνεται και η υποβολή παραπώνων. Το να περιληφθεί σε άλλη οδηγία δεν σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια. Γι' αυτό θα ζητήσω από την ε, πολιτική μου ομάδα να μην υποστηρίξει αυτή την πρότασή του συγητού. να ζητήσω και από την, πάλι από την πολιτική ομάδα να καταψηφίσει ορισμένε τροπολογίε του εισηγητού. Διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή πέραν των ευθυνών τη ε, χώρα τη σημαία. Διότι ευθύνη φέρει η χώρα ε, της σημαίας για να επιβάλλει τις διατάξεις της οδηγίας 2009-13 και αναμένω την ψηφοφορία. Η πρόεδρος, Επιθυμεί άλλος κανείς να λάβει το λόγο. Υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ναι, εσείς. Λέγομαι Μπέρκ από την DG Move. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. υπήρξε μείζον δυστύχημα χθες το βράδυ και εκφράζουμε τη λύπη μας ένα μεγάλο σκάφος μεταφοράς οχημάτων συγκρούστηκε με άλλο σκάφος 69 μίλια έξω από το Ρότερνταμ. Δυστυχώς σε αυτή την ε, ώρα έχουμε ακόμα 7 αγνοωμένους οι επιχειρήσεις διασώσεως γίνονται από τις ε, λιμενικές αρχές. Διασώθηκαν 13 μέλη του πληρώματος μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα λόγω των συνθήκων, των θαλάσσιων συνθήκων εκεί, δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να ε, μπορούν να διασωθούν οι 7 Και οι σκέψεις μας και οι σκέψεις του Επιτρόπου μας Κάλλας ε, είναι βεβαίως με τις οικογένειες των αγνωμένων και των, και των, ε, και των ε, ναυαγών. Βεβαίως ατυχήματα συμβαίνουν. Αυτό ρίχνει ένα ιδιαίτερο φως σε πολλές από τις συνθήκες που πρέπει να παρακολουθούνται όταν ναυσιπλοεί κανείς και οι συνθήκες εργασίας βέβαια είναι σημαντικό στοιχείο. Θεωρούμε λοιπόν ότι το συμπέρασμα μάλλον η ολοκλήρωση, η ολοκλήρωση του πακέτου του 2006 για την ναυτική εργασία και η συμφωνία που επέτυχαν οι κοινωνικοί εταίροι που έχει περιληφθεί στην οδηγία 2019-2013 είναι σημαντικά και γι' αυτό η Κομισιόν προσπαθεί τώρα ε, να περάσει τις διατάξεις έγκαιρα για τις ευθύνες των χωρών της σημαίας ώστε <clears throat> να είναι έτοιμες όταν θα ισχύσει και η συνθήκη του χρόνου, το επόμενο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει τα μέλη σας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στην προσέγγιση. Η Κομισιόν έχει προσπαθήσει να επιβάλλει το περιεχόμενο της συμφωνίας. Σημείωσα το περιεχόμενο της δηλώσεως που ανέγνωσε ο σκιώδης Εάν θεωρείτε, κυρία Πρόεδρε, ότι όλον το κείμενο της MLC πρέπει να είναι αναγκαστό, η Κομισιόν δεν αντιτίθεται εξ αρχής, αλλά βέβαια θα πρέπει αυτό να γίνει αντικείμενο συνεννόησης για να βρεθεί συμφωνία με τον συνομοθέτη, το Συμβούλιο. Σημειώνουμε ωστόσο ότι υπάρχει ένας αριθμός στοιχείων στην MLC που θα είναι δύσκολο να μπορέσουν να περιβληθούν τον μανδύα των εφαρμοστικών διατάξεων, ιδίως για ορισμένες υπηρεσίες που επιφέρουν ένα στοιχείο εξοδαφικότητας του α, κοινοτικού νόμου, διότι οι συμβάσεις εργασίας πληρωμάτων ή μελών πληρωμάτων μπορεί να αναφέρονται, να παραπέμπουν δηλαδή είτε στην χώρα της σημαία ή του ship manager ή και της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα, όπου κατοικεί δηλαδή ο ναυτικός. Πρέπει να δούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι με ποιο μέσο ή με ποια μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να επιβάλλει την εφαρμογή της MLC από τις ενδεχόμενες τρίτες χώρες οι οποίες εμπλέκονται. Εμείς οι ίδιοι είμαστε διατεθειμένοι να αρχίσουμε να το εξετάζουμε ένα ε, σύστημα ίσως πιστοποίησης και επιθεώρησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας καθώς επίσης και από την ε, άποψη της εκπαίδευσης και υπό την, ε, υπό την Σύμβαση STC να πηγαίνει η Maritime Agency να διοργανώνει εκπαιδεύσεις και σε τρίτες χώρες για πληρώματα που θα εργάζονται σε ευρωπαϊκά πλοία. Βέβαια αυτό είναι μέγα εγχείρημα και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρήσαμε ότι έχει οριμάσει τέτοια πρόταση. Και επίσης υποχρώσεις των, του, της χώρας του Λιμένα και της σημαίας να διατηρηθούν και ενδεχομένως να εξετάσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι κατάλληλο για να επιβληθεί εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Υπάρχει πολύ καλή θέληση με την οποία συμφωνούμε στην πρότασή σας. Είναι όμως δύσκολο και ακαθόδες το θέμα σε ό,τι αφορά την εξοδαφική εφαρμογή. Και από την πλευρά της Κομισιόν ε, θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για τη σχετική μελέτη. Και το άλλο κύριο θέμα που θέλω να θέσω είναι για μια ενδεχόμενη διπλή πιστοποίηση όπου δεν βλέπουμε να προκύπτει ευεργέτημα υπέρ των χωρών μελών να εκδίδουν δηλαδή πρόσθετα πιστοποιητικά που να σχετίζονται με την οδηγία 2009-13 γνωρίζοντας ότι σε ό,τι αφορά ισότιμο ανταγωνισμό ο έλεγχος του τελικού λιμένα θα πρέπει ε, με αυτόν τον τρόπο να γίνονται οι έλεγχοι όλων των σκαφών που ε, έρχονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και να εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Για πολλές από τις τροπολογίες έχουμε την πεποίθηση ότι στη συνεργασία μαζί σας αλλά και με το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε διατυπώσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την ταχεία πρόθεση της ε, συμφωνίας για την εφαρμογή της οδηγίας που είναι σημαντικό στοιχείο και που θα πρέπει να είναι όπως είπα ήδη ε, να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ όταν θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη το επόμενο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ καθώς επίσης ευχαριστώ και για την συνεργασία όλα τα μέλη σας. Ευχαριστώ για τα στοιχεία που θέσατε υπόψη μας λέει η Πρόεδρος διότι δείχνει το δυναμισμό ε, του θέματος και του κειμένου και επιτρέπει να ανοιχθούν κάποιοι δρόμοι για να σημειωθεί πρόοδος με πιο ικανοποιητικό τρόπο αντί απλώς να γίνει μονάχα η μεταφορά της Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων. Είναι σημαντικό βέβαια αυτό, αλλά πριν από την θέση ισχύ της συνθήκης. Από την άλλη μεριά σε αυτήν την προσπάθεια των μικρών βημάτων λησμονούμε ε, τα θεμελιώδη που είναι η συνθήκη, η σύμβαση για την ναυτική εργασία με συνεργασία και των, τρι, και των τρίτων χωρών που γνωρίζουμε ότι αυτές είναι κέριο θέμα. Νομίζω ότι αναφέρατε και το ναυτικό δράμα που ε, συνέβη χθε τη νύχτα. Ποιε σημαίε έφεραν τα σκάφη αυτά και ποια ήταν η κατάσταση των πληρωμάτων. Πράγματι, απάντηση της Κομισιόν. Αφενός ήταν ένα σκάφος με βοημική σημαία ε, μεταφοράς οχημάτων, βαλτικής χώρας δηλαδή, με φορτίο 1.400 νέων καινούριων αυτοκινήτων, με πλήρωμα 24 μελών, από τα οποία διασώθηκαν τα 13 και 7 αγνοούνται και 4 δυστυχώς ανεβρέθησαν νεκροί. Και από την άλλη ένα σκάφος με κυπριακή σημαία, κόλβους J, όλα τα μέλη του πληρώματος αυτού του σκάφους είναι ΣΟΑ και συμμετέσχουν ενεργώς στην επιχείρηση διασώσεως το σκάφος αυτό ήταν μικρό εμπορευματο... Ε, ε, ε, σκάφος εμπορευματοκιβωτίων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, διευκρινήσεις αυτές. Άλλο ένα ναυτικό δράμα. Στις 12 Δεκεμβρίου προβλέπεται συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές. Θα δούμε πώς θα περιλάβουμε τα διάφορα αυτά στοιχεία έχοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετάσουμε τις ενδεχόμενες τροπολογίες συμβασμού μέχρι τις 23 Ιανουαρίου και να ψηφίσουμε στις 24 Ιανουαρίου ώστε να καταλήξει το κείμενο στην Ολομέλεια ενδεχομένως Μάρτιο-Απρίλιο εκτός αν προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Τελειώσαμε αυτό το θέμα της ημερησίας διατάξεως και... και... περνάμε στο σημείο 13 κοινή συζήτηση των δύο εκθέσεων του κυρίου Χόουιτ προβλέπεται στο σημείο αυτό αλλά απουσιάζει ο κύριος Χόουιτ Σας πειράζει να εξετάσουμε πρώτα το σημείο 15 της κυρίας Όμεν Ρόιτον που είναι παρούσα. Για να δούμε, είναι εδώ οι σκιώδεις ηγητές. Μα δυστυχώς δεν βλέπω να είναι παρόντες όλοι οι σκιώδεις ηγητές για το 15. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος, ο κύριος Χόουιτ ή και ο για το 15. Ε, δυστυχώς πρέπει να επιστρέψω, γιατί έχει ένα πρόβλημα η μητέρα μου και να φύγω το συντομότερο δυνατό. Μπορούμε να καλέσουμε τους και οδησηγητές. Ναι, ε, ναι. Είπα ότι μάλλον το δικό σας θέμα θα συζητηθεί πριν το θέμα του κυρίου Χόουιτ. Όλοι έχουμε υποχρεώσεις, φυσικά έχουμε κατανόηση και για τις δικές σας. Να δούμε αν είναι παρούσες οι διαπραγματευτικές ομάδες, οι σκιώδεις ηγητές και για τα δύο θέματα. Ensemble des interlocuteurs, donc je ne pense pas que c'est de bonnes euh, pratiques. Voilà, mais on, τι μας ε, προτείνετε κύριε Σέρκας. Όντως, απουσιάζει ο σκέδης ηγετής μας, τον φωνάξαμε. Αλλά από τη στιγμή που έχει πρόβλημα κυρία κυρία ήταν ε, ας ξεκινήσει και θα σημειώσω εγώ τις παρατηρήσεις για να τις διαβιβάσω στο σκιώδη ηγετή μας αλλά ακόμη και δεν έρθει ο σκιώδης συγκεκριτής, μπορώ εγώ να μεταφέρω κάποιες ε, σκέψεις των σοσιαλιστών. Bien, il est 11h35. Euh, nous... Είναι 11 και 35. που είχαμε προγραμματίσει για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Οπότε, μια και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ποιος ήρθε? Ο κύριος Δαρντέν πρόλαβε ή ο κύριος Χόβιτ. Α, ο κύριος Δαρντέν, θαυμάσια. Οπότε, θα περάσουμε στο σημείο 15, έκθεση ο Ρόιτεν. γιατί δεν βλέπω να έχουν αντιρρήσει ούτε οι πράσινοι ούτε οι φιλελεύθεροι. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας λοιπόν, την κυρία Όμεν Ρόιτεν, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής της με θέμα το πρόγραμμα για τις επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Φεβρουαρίου είχε δημοσιεύσει τη Λευκή Βίβλο της και η έκθεσή μας αποτελεί αντίδραση ως προς την δημοσίευση αυτή. Όπως είπε κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς πήγαμε να φύγω το συντομότερο δυνατό. Η μητέρα μου έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να σπεύσω λοιπόν ε, και να φροντίσω να μεταφερθεί με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Κύριε Πρόεδρε. Om ook de toelichting goed te lezen, omdat hij precies, denk ik. Οι συνάδελφοι ελπίζω να διάβασαν την αιτιολογική έκθεση γιατί παρουσιάζει πιστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα κράτη-μέλη. Εγώ βέβαια είμαι Ολλανδέζα, αλλά προσπάθησα στην έκθεσή μου να καλύψω την κατάσταση όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα αφορούν εθνική αρμοδιότητα. Υπάρχει όμως ανάγκη πανευρωπαϊκού συντονισμού. Και όταν βλέπουμε τους όρους της συνθήκης, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη στρατηγική το 2020, δεν μπορούμε παρά να κρίνουμε ότι θέματα συντονισμού είναι η καλύτερη περίπτωση και ένας τρόπος soft law, μη δεσμευτικού δικαίου για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη συνεννόηση. Δυστυχώ λόγω της ενεργείας, ο κόσμος αρχίζει και δουλεύει όλο και πιο αργά, βρίσκει δουλειά όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία Ik hoop Ελπίζω να τα καταφέρω τώρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Οι νέοι παρόλο που είναι ειδικευμένοι και έχουν πολλά προσόντα δεν βρίσκουν δουλειά. Μπαίνουν στην αγορά εργασία πολύ αργότερα. Ενώ ταυτόχρονα επιμηκύνουμε την ηλικία συνταξιοδότηση. Μειώνεται λοιπόν ε, το, ο ενεργός πληθυσμός και το 2008 ε, είχαμε τέσσερις εργαζόμενους που πλήρωνε φορές για ένα συνταξιούχο, ενώ το 2020 αναμένεται ότι θα έχουμε πολύ χειρότερη κατάσταση. Αν δούμε πόσο ο κόσμος το 1960, είχαμε προσδόκιμο 67 χρόνια για τους άνδρες ενώ το 2004 είναι 76 το προσδόκιμο ε, για τους άνδρες και 82 για τις γυναίκες. Αλλά είναι και χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, και με μεγάλες διαφορές φυσικά μεταξύ των χωρών μελών. Στις κάτω χώρες, ε, οι άνω των 55, οι άνω των 55, θα είναι σε 53%, ενώ στη Σουηδία 73%. στη Δανία 61% και στο Βέλγιο 31%. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν σε προχωρημένη ηλικία με καλή υγεία και άρα εξαρτώνται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Δεδομένων στη συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, δεν υπάρχουν ε, άνθρωποι που να εργάζονται, που να πληρώνουν ε, τις ε, εισφορές τους, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι συντάξεις. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα παρουσιάζουμε εδώ. Υπάρχουν βέβαια διάφορα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, ισχύει το πιο κοινό και σημαντικό σύστημα που είναι το σύστημα του πρώτου πυλώνα με βάση το οποίο η πληρωμή των συντάξεων γίνεται μέσω χρηματοδοτή από τις κοινωνικές ε, παροχές, από τις εισφορές και τις φόρους. Αλλά δυστυχώς οι, οι συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν αυξάνονται λόγω της αύξησης των συνταξιούχων και απορροφούν μεγάλο τμήμα του προπολογισμού. Τι κάνουν τότε τα κράτη. Είτε συσσωρεύουν δημοσιονομικό έλλειμμα, κάτι που απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή καλούνται να περικόψουν τις πληρωμές. Οι συνταξιούχοι μας όμως χρειάζονται ένα ξεπρεπές εισόδημα για να επιβιώσουν. Γιατί ειδικά τους συνταξιούχους πλήττει το φαινόμενο της φτώχειας. Δεν θέλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Θέλουμε αξιοπρεπείς συντάξεις αλλά και η υγιή οικονομική κατάσταση των χωρών μελών και δημοσιονομική εξυγίαση. Θα πρέπει λοιπόν με τα συστήματα που θα θεσπίσουμε και να κάνουμε κάποιες οικονομίες και να δούμε ποιος πυλώνας θα επηρεάζεται από τις περικοπές, ο πρώτος ή ο δεύτερος. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε και εμπράκτος την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και μάλιστα σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Βέβαια δεν μπορεί όλη αυτή η πίεση να βαρύνει τους νέους που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας. Ανέλησα λοιπόν την κατάσταση και υπέβαλα κάποιες προτάσεις. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, θέσεις απασχόλησης για όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας γιατί είναι απαράδεκτο ενήλικοι άνω των 55 να είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης και των απολύσεων, ακριβώς επειδή είναι ακριβή για τους εργοδότες. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές, ώστε και οι ενήλικες άνω των 55 που θέλουν να συνεχίσουν να απασχολούνται, να μπορούν να κρατήσουν τη δουλειά τους και με κατάλληλες αποδοχές. Η κατάσταση βέβαια διαφέρει, όπως σας είπα, από χώρα σε χώρα και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν οικονομίες, άσχετα με το συνταξιοδοτικό σύστημα που εφαρμόζεται. Θα πρέπει να γίνουν οικονομίες και στον πρώτο, αλλά και στο δεύτερο πυλώνα. Και πιστεύω ότι άσχετα με το σύστημα που θα επιλέξουμε, τα το βασικό του χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι η ασφάλεια. Και γίνονται επενδύσεις στο δεύτερο πυλώνα και στα συνταξιδοτικά ταμεία που τα διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητούμε έντονα δηλαδή οι επενδύσεις των συνταξιδοτικών ταμείων είναι βιώσιμες. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνουν σχετικές προσαρμογές στην ε, οδηγία. Και οι απαιτήσει ε, φερεγγιότητας να περιλαμβάνονται στην οδηγία IORP. Εγώ είμαι αρκετά επικριτική για το θέμα αυτό. Και περνάω στο επόμενο θέμα, την ενημέρωση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενημέρωση. ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι γιατί τους για το τι θα τους περιμένει όταν θα βγουν στη σύνταξη. Θα πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν. Και αν θέλουν σύνταξη θα πρέπει να καταβάλουν τις φορές τους. Επίσης, το θέμα της κινητικότητας είναι πολύ σημαντικό. Πέρσι, στη Πράσινη Βίβλο, είπαμε ότι δεν θα πρέπει να διακυβεύεται κινητικότητα. Και αυτή είναι μια πρόταση που απασχόλησε ιδιαίτερα την Κυπριακή Προεδρία. Γιατί δικαίωμα για σύνταξη έχουν όχι μόνο οι στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο πυλώνα. Και θα πρέπει να υποφελούνται από αυτό το σύστημα ακόμη και αν χρησιμοποιούν ε, την κινητικότητα. θα πρέπει κανείς να μπορεί να μεταφέρει το κεφαλαίο του όταν μετακινείται. Αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε και σε κάποιες ελάχιστες συμφωνίες ε, για τα δικαιώματα, τα συνταξιοδοτικά. γιατί οι άνθρωποι κάνουν οικονομίες, επενδύουν στα, στα εξοδοτικά τους ε, συστήματα, θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται λοιπόν μια βιώσιμη σύνταξη. Και ίσως ο κανονισμός 883 μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλά προσοχή μην χαθούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε μια πρόταση υπερβολικά διεξοδική και δεν ξέρω αν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό συνταξιδοτικό ταμείο για τους ερευνητές. Εγώ δεν βλέπω τη σκοπιμότητα μιας τέτοια πρότασης, αλλά περιμένω και τη γνώμη των συναδέλφων. Κοντολογής. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών, θα πρέπει να εφαρμόσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Εγώ σκιαγράφησε κάποιες μεταρρυθμίσεις και σε ό,τι φορά την οδηγία IOPR είπε ότι έχω αρκετές επιφυλάξεις αλλά είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής για τις ποσοτικές απαιτήσει. Τώρα αν μιλούμε για ποιοτικέ απαιτήσει, δηλαδή χρηστή διαχείριση, ε, διακυβέρνηση και διαφάνεια των συνταξιδοτικών ταμείων, ε, με αυτά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αυτά ζητώ συγγνώμη γιατί τα προσωπικά μου προβλήματα μου δημιούργησαν μια νευρικότητα. Έχασα τη φωνή μου λόγω το βήχα, αλλά αυτά οφείλονται στο άγχος που έχω και στην ανησυχία μου για τη μητέρα μου. Ε, ευχαριστούμε συνάδελφε, αγαπητοί συνάδελφε. Οι σκιώδες εισηγητές δεν είναι εδώ, μόνο ο κύριος Νταρντέν και ο κύριος Ντεμπάκερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια γιατί είμαστε στην αρχή αυτής της σημαντικής συζήτησης και αυτής στην πρώτη ανάλυση και θα ξανασυζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και εκ νέου με την κυρία Όμεν Ράιτον όπως κάναμε και για το πράσινο βιβλίο. Σημαντικό θέμα το λέγαμε και για το πράσινο βιβλίο ότι δηλαδή σε επίπεδο κρατών μελών και εθνικών προϋπολογισμών η κατάσταση είναι ε, δύσκολη και η πτυχή σύνταξη είναι ένα σημαντικό θέμα. Τα περιθώρια λιγμού είναι μικρά Πρέπει να σκεφτούμε το θέμα αυτό με όλα αυτά στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε μόνο προϊόν τους προϋπολογισμούς, μόνο τα χρήματα. Πρέπει <clears throat> να έχουμε υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης που θα πρέπει να παραμείνει στην βάση αυτού του συστήματος του εξαιρετικού και οι πολίτες το χρειάζονται. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει στην έκθεσή μας και στον προβληματισμό μας και μάλιστα σε μια στιγμή όπου η επισφάλεια όλο ένα και αυξάνεται. Τώρα έχουμε την ετήσια σύμβαση του της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της στόχης και δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι αντί να βλέπουμε τον αριθμό των ανθρώπων, των φτωχών ε, να μειώνεται, βλέπουμε και διαπιστώνουμε το αντίθετο. Άρα τα συστήματα τα συνταξιδοτικά θα πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της στόχιας. Και το μέλλον των συντάξεων είναι μια μεγάλη πρόκληση. Στο πλαίσιο του πράσινου βιβλίου και μπορώ ήδη να το πω και να το επαναλάβω, οι βασικές γραμμές είναι η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις σημαντικές τους πυλωτικούς πυλώνες της αλληλεγγύης ε, να έχουμε όχι μόνο την αύξηση του νόμου ηλικίας δεξιδότησης αλλά θα πρέπει και εδώ να δώσουμε αποχρώσεις ανάλογα με τα κράτη-μέλη γιατί τα συστήματα είναι πολύ διαφορετικά από το ένα μέρος στο άλλο και πολλές φορές και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται δεν σημαίνουν το ίδιο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχυση. Το ταμείο, το συνδεξιωτικό μπορεί να συνδέεται με τον ένα πυλώνα ή τον δύο πυλώνα σε κάθε χώρα. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε την κινητικότητα των κανόνων που ισχύουν, των κανόνων πρόνοιας. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και εδώ, γιατί δεν θα πρέπει να εξισωθούν υπερβολικά αυτά τα ταμεία με άλλα είδη ταμείων πιο κερδοσκοπικών. Ε, αυτά είναι κάποια στοιχεία για τα οποία θα επανέλθουμε. Και για το σχέδιο το οποίο εσείς συντάξατε, νομίζω πως υπάρχουν πολλά πράγματα ενδιαφέροντα εδώ. Να φτάσουμε στο να διαβάσουμε την συμβιβαστική. Έχουν εδώ υπάρξει κάποιες ετοιμήσεις για θα πρέπει να τα ξαναδούμε γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς εγώ αυτό ως συμβιβαστική. Πάντως εν γέννη αποκατάσταση της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης ε, το ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται ακόμα και αν είναι ηλικιωμένοι και να υπάρχουν δεσμοί ανάμεσα σε διάφορους εργαζόμενους οι διάφορες πτυχές όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Κύριε, ο κύριος Δεμπάκερ και μετά ο Τόμας Μαν που είναι εισηγητής για αυτό το λευκό βιβλίο. Κύριε Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Την εισηγήτρια, με συγχωρείτε. Ε, επίσης ε, ήταν πολύ καλό που μπορέσαμε, μπορούμε να συζητήσουμε την άποψή μας για το λευκό βιβλίο. Αν λάβουμε υπόψη κάποιους ε, παράγοντες όπως η, η γύραση του πληθυσμού, η δημοσιονομική περιορισμή των κρατών μελών, νομίζω πως έχουμε να κάνουμε με το πιο σημαντικό και επίγοντα φάκελο για τους πολίτες αυτή τη στιγμή σε αυτή την Επιτροπή. Για τις συντάξεις βεβαίως βασική και κεντρική ευθύνη βαραίνει τα κρατη Είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια εκτίμηση για το ποια είναι η κατάσταση των διαφόρων συνταξιδοτικών συστημάτων στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση. Να δουλέψουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκή βάση και να εγγυηθούμε και κάποιες πτυχές κινητικότητας και αλληλεγγύης για τις οποίες ήδη μιλήσαμε. Ο εισηγητής επίσης αναφέρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απασχόληση και την σύνταξη και αυτό θα έπρεπε να είναι ευρύτερο με την έννοια ότι σήμερα βλέπουμε πολλές σύγχρονες, πολλές σύγχρονες σύγχρονες μορφές εργασίας, σχήματα εργασίας που δεν καλύπτονται από τα στεξιδοτικά ε, ταμεία όπως τα είχαν ε, καλυφθεί παλιότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη και να τονίσουμε πως οι ίδιοι οι απασχολούμενοι έχουν δικαίωμα σε μάξιμο ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα και μάξιμο ε, συνταξιδοτικών ε, δικαιωμάτων. Είμαι υπέρ λοιπόν αυτής της δικαιοσύνης που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συζητήσεις μας. Ε, συμφωνώ επίσης ότι πολλές ε, ε, από τις συντάξεις θα πρέπει να είναι βιώσιμες, να υπάρχουν δηλαδή συστήματα και να μπορέσουν να προσαρμοστούν και τα συνταξιδικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες και σε συλλογικό και σε μεμονωμένο επίπεδο γιατί ένα συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε προς ένα ε, καλύτερο σύστημα. Ε, Επίση, έχουμε δύο αλλαγέ στο δημοσιονομικό κανονισμό. Έχει ενισχυθεί πολύ αυτό ο κανονισμό και επί τη βάση τη στήριξη αυτή ε, το στηρίζουμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην προκαλέσουμε μη επιθυμητέ επιπτώσεις που δεν θέλουμε ε, γιατί σε κάποια κάτι μέλη λειτουργούν τα πράγματα και μπορεί τελικά να καταλήξουμε σε υπερρύθμιση. Να προσέξουμε πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ ε, σπουδαίο σύστημα και πρέπει να εξασφαλίσουμε την ορθή του λειτουργία. Να προσέξουμε και την ε, συνειδητοποίηση και την κατάρτιση του κόσμου. Γιατί οι προσδοκίες του κόσμου δεν είναι αντίστοιχες με την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε με διαφανή και ακριβή τρόπο. Και ε, πολλά κράτη-μέλη που έχουν φτιάξει υπηρεσίες για να παρακολουθούν την εξέλιξη των συντάξεων ε, ε, βοηθούν, βοηθούν τους πολίτες ώστε να έχουν μια σωστή αξιολόγηση για το, για το τι θα έχουν να λαβαίνουν στο μέλλον. Κάποια στοιχεία ακόμα πρέπει να συζητηθούν, να αναφέραμε πως είναι μια αξιόπιστη ε, κατάσταση. Ειδικά στο Βέλγιο βλέπουμε πως οι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, ε, ας πούμε στο Βέλγιο λειτουργούν ε, στο δεύτερο πυλώνα και παρέχουν και μακροπρόθεσμη βοήθεια και σύνταξη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Να λάβουμε υπόψη δηλαδή την ιδιαιτερότητα των κρατών μελών. Πολύ αξονικό σύστημα δηλαδή επικρατεί δεν είναι εύκολο να συνδυαστεί με τη σημερινή πραγματικότητα γιατί μπορεί οι εργοδότες να μην, να μην είναι σε θέση να συμβάλλουν λόγω των οικονομικών δυσχερίων. Έχουμε και άλλες παρατηρήσεις, αλλά ε, θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο Τόμας Μαν και μετά ακολουθούν πέντε, δηλαδή τέσσερις μάλλον, Παρακαλώ λοιπόν όλες και όλους να μείνετε μέσα σε κάποια χρονικά όρια. Τόμας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατάλαβα ότι έχω περιορισμένο χρόνο και θα το σεβαστώ με την Ρία Όμεν, στο πρόσωπο μάλλον Ρία Όμεν, ε, έχουμε μια εξαιρετική εισηγήτρια την οποία γνωρίζουμε και από παλαιότερα. Ρία, δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει όλα, αλλά μπορεί κανείς να ψηφίσει και να ε, εγκρίνει ε, ορισμένες βασικές αρχές, κυρίως ό,τι αφορά την δυνατότητα χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων για το μέλλον. Πριν ε, από λίγο ήμουν στους πρώην ευρωβουλευτές που είναι συνταξιούχοι τώρα και οι οποίοι παρακολουθούν προσεκτικά τις συζητήσεις μας και βλέπω ότι και οι απόψεις τους είναι πολύ ενθαρρυντικές. Για τον πρώτο ή δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να συμπληρωθεί είναι σωστό αυτό. Ορισμένες χώρες μέλη όμως αμφισβητούν τους πυλώνες και μιλούν για τρίτο πυλώνα. Με, κάθε, με όλες τις διαφορές τις οποίες έχουμε πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε πώς, δεν θα, πώς θα αποφύγουμε ένα άκαμπτο σύστημα το οποίο να μην επιτρέπει τη χρηματοδότηση των συντάξεων από επιχειρήσεις. Εγώ τα έχουμε συζητήσει και με τα θέματα Solvency και η στην Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Απασχολήσεως και η Οικονομική Επιτροπή ασφαλώς θα καταλήξουν σε κάποια κοινά θέματα. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Γερμανία θέλουμε, λέμε ότι θέλουμε να αμείβονται αυτοί οι οποίοι παραμένουν πιστοί στις επιχειρήσεις, αυτοί δηλαδή οι οποίοι εργάζονται σε μια επιχείρηση πολλά χρόνια, να πάρουν ένα είδος μπόνους. Αυτό δεν σημαίνει όπως λένε ορισμένοι περιορισμό της κινητικότητας, η κινητικότητα βεβαίω δεν πρέπει να τιμωρείται, σωστό, αλλά δεν είναι φρένο στην κινητικότητα για εκείνους οι οποίοι είναι δεχτοί στις επιχειρήσεις ε, να πληρώνονται οι ε, συντάξεις από τι επιχειρήσεις. Ρία, είναι σωστό που λε ότι οι κρατήσεις για συντάξεις από επιχειρήσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το δούμε. Έχουμε λοιπόν κοινέ αρμοδιότητε και στι δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, Έχουμε και άλλε αρμοδιότητε, Εγώ σα θα πω το εξή, κυρία Πρόεδρε, λόγω τη συζητήσεω που είχα πριν λίγο στην Οικονομική Επιτροπή όταν εδώ διεξήγεται η ε, ε, ψηφοφορία σε εσά, είχα την έκθεσή μου στην Οικονομική Επιτροπή, τέθηκαν πολλέ ερωτήσει, οι οποίε στην πραγματικότητα είναι και αρμοδιότητα δική μα εδώ. ορισμένε από τι τροπολογίε που θα ε, ε, υποβληθούν εκεί, μπορούμε σίγουρα να τις εξετάσουμε και εδώ, γιατί έχουμε και θέλουμε να έχουμε πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο εκθέσεων. Αυτά πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Καλά λοιπόν, ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι αγορητές, ο κύριος Όρη πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω και λίγα λόγια ε, υπό την προσωπική μου ιδιότητα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Χαίρομαι για την έκθεση και ευχαριστώ ιδιαίτερο στην Ρία Όμεν. Πρόκειται για μια έκθεση πραγματικά ισορροπημένη η οποία λαμβάνει υπόψη πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει στην παρούσα Επιτροπή. Η Ρία Όμεν μιλεί για την ευθύνη των επιμέρους χωρών και εξετάζει τα συνταξιωτικά συστήματα όχι σαν ένα οποιοδήποτε οικονομικό προϊόν ή επιχείρηση ή σαν ένα, σαν ένα οικονομικό πρόβλημα. Η, η κοινωνική αλληλεγγύη και τα συστήματα κοινωνική αλληλεγγύη είναι ζήτημα ευθύνη των χωρών μελών. Η κυρία Ρία Όμερ μιλεί και για την κινητικότητα. Σωστό. Μπορούμε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο με ποιο τρόπο και με ποια μέσα θα ενισχυθεί η κινητικότητα. Κάτι που ε, νομίζω λείπει είναι το εξή. Μιλούμε και σε άλλα πλαίσια συχνά για το ότι μετά από την παρούσα κρίση τίποτε πλέον δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν. Αυτό το είπαμε ήδη σε σχέση με την δομή της απασχόλησης, τη διάρκεια των ε, συμβάσεων εργασίας. Δεν βλέπω εδώ να περιλαμβάνεται τίποτε σχετικό με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν νέες μορφές απασχολήσεως, άτυπες μορφές απασχολήσεως, νέες μορφές συμβάσεων και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται νέες μορφές αυτές πρέπει να τις ε, συμπεριλάβουμε, να τις διοχετεύσουμε, να ενταχθούν και αυτές στα συνταξιωτικά, συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να μνημονευθούν στην έκθεση. Υπάρχει και ένα θέμα στο οποίο ε, έχω άλλη άποψη από την εισηγητρία σε σχέση δηλαδή με τον δεύτερο πυλώνα. Εκεί διαμορφώνονται διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν χώρες μέλη δηλαδή όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην οικονομία και άλλες όπου κυριαρχούν περισσότερο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, επιθυμείτε να τελειώσω. Είναι σωστό που η Ρία τα θίγει τα θέματα αυτά. Αλλά εν τέλει πρέπει όλοι να δουλέψουμε περισσότερο και πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να δουλέψουν περισσότερο. Η απασχόληση είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούτα Στάινρουκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλές είναι οι προθέσεις, θετικές, ωστόσο οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε στην, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να οδηγούν μονάχα σε περικοπές των κοινωνικών συστημάτων που θίγουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα εξαρτώνται αργότερα από την σύνταξη. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της σύνταξης αλληλεγγύης. Χρειάζεται επίσης να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε κατά της φτώχειας των γυρατιών. Διαβάζω στην πρόταση της Κομισιόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ιδιωτικές συντάξεις. Άνθρωποι οι οποίοι ε, κερδίζουν λίγα ή δεν έχουν καν ε, απασχόληση, έχουν άλλα προβλήματα. Πώς θα χρηματοδοτήσουν και την ιδιωτική ε, ασφάλιση, ιδιωτική σύνταξη. Υπάρχουν και εθνικές ιδιαιτερότητες. Σωστό, το είπε και ο κ. Μαν. Στη Γερμανία ο δεύτερος πυλώνας με την, συνθήκη, με την ε, ε, σύνταξη μάλλον από επιχειρήσεις είναι εθελοντικός, δεν είναι προϊόν, δεν είναι οικονομικό προϊόν, είναι καθαρά πρόνοια. Οι προτάσεις τη Κομισιόν θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με 50 περίπου δις ευρώ. Αυτό θα σημαίνει τον θάνατο του δεύτερου πυλώνα. Δύο τρίτα των εργαζομένων λαμβάνουν συντάξεις από τις επιχειρήσεις αυτές. Και μέχρι 50% λαμβάνουν τις ε, συντάξεις τους. Είναι το 50% των συντάξεων το λιγότερο. Αυτό. Να μην καταστραφεί αυτός ο δεύτερος πυλώνας. Αλλά η καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης τη φτώχειας των ηλικιωμένων είναι να οι άνθρωποι να έχουν δουλειά και να αμείβονται καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτριά μας. Αυτά που είπε το Κοινοβούλιο για την Πράσινη Βίβλο εισακούστηκα στη Λευκή Βίβλο ή πήγαν τελείως χαμένες στο Ρόντο οι παρατηρήσεις μας. Τις έλαβε καθόλου υπόψη τη Λευκή Βιβλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε υπάρχει και μια παλιά ιδέα λέω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουμε την κινητικότητα αλλά και ότι αυτοί έχουν δικαίωμα για ένα 28ο, ένα συνταξιδικό καθεστώ διαφορετικό από αυτό που ισχύει στι 27 χώρε μέλη. Είχα καταλάβει στην αρχή της κοινοβουλευτικής μας θητείας όταν ανέλαβα την Προεδρία ότι μας έμεινε και το θέμα της ε, μεταβασιμότητας ε, των ε, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια πράσινη βίβλο, θα έδινε μια μαγική λύση για όλα αυτά. Βέβαια, έχουμε ήδη τη λευκή βίβλο και δεν βλέπω να έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Τι γίνεται ε, υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης των συνταξιδοτικών ε, δικαιωμάτων. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση των εθνικών ε, συνταξιδοτικών μοντέλων. Και δεν μπορούμε φαινώς να ενισχύουμε τα εθνικά αισθήματα και ταυτόχρονα ε, την μεγάλη κινητικότητα από τις περιφερειακές χώρες, γιατί εξαιτίας της κρίσης το θέμα της ισότητας ε, στα δικαιώματα και στην εργασία είναι ένα θέμα που ξαναβγαίνει στο προσκήνιο με το οικονομικό μοντέλο και οι, εργαζόμενοι και οι πολίτες από την περιφέρεια προτιμούν ε, να εργάζονται σε μια χώρα του κέντρου και να επιστρέφουν για την ε, σύνταξή τους στις πατρίδες τους. Το θέμα λοιπόν της τη δυνατότητα μεταβίβασης ε, των ε, συνταξιδοτικών δικαιωμάτων θα πρέπει να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα και να το ευθαγραμμίσουμε με τις νέες συνθήκες και εξελίξεις και την νέα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Ελπίζω όλα αυτά να βρουν μια αντανάκλαση στην έκθεση. Κυρία Γεζοβιέτσκα. Έφυγε. Κύριε Κορνέλισεν. <laughs> Sorry, I thought that was somebody συγγνώμη, νόμιζα ότι προηγούνταν άλλος συνάδελφος. Μα γι' αυτό μιλούσε για τους μετανάστες, την εσωτερική μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ την εισηγητρία, πολύ ισορροπημένη η έκθεσή τη. και πολύ καλό σημείο εκκίνησης και βάση για τη δουλειά μας. Λέμε ότι χρειαζόμαστε μία μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση ενώ δυστυχώς τα κράτη-μέλη επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμες πολιτικές συλλητότητας και αποσπά την προσοχή τους από την ανάγκη πιο μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων. Η έκθεση ε, δίνοντα, ε, ξεκινά δίνοντας έμφαση στον κίνδυνο της φτώχειας ε, για τους ηλικιωμένους, τεράστιος κίνδυνος και απειλή και είναι ακόμη πιο τρομακτική γιατί δυστυχώς αυτοί που έχουν μπει στη σε καθεστώς ε, συνταξιοδότηση δεν μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασία και οπότε δεν μπορούν να, να αποσοβήσουν αυτό το φάσμα τη φτώχειας. Ε, υπάρχει ανάγκη εξασφάλιση και του ελάχιστου αξιοπρεπού εισοδήματο για τους συνταξιούχου, να το τονίσουμε και αυτό. Κάτι που λείπει ίσω από την έκθεση είναι η συντάξει για τις ιδιαίτερα ευάλωτε ομάδε, όπω είναι οι γυναίκε που αποφελούνται από την άδεια μητρότητας ε, ή από μετανάστες που ακριβώς επειδή μεταναστεύουν και εργάζονται σε προχωρημένη ηλικία δεν έχουν πια έχουν χάσει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, έχουν ελάχιστα στη χώρα τους. Να μην ξεχάσουμε και αυτές τις κατηγορίες των πιο ευάλωτων εργαζομένων. Στην παράγραφο 14 είναι σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη αλληλεγγύης γιατί σίγουρα οι συντάξει είναι άσκηση αλληλεγγύης και αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να το διαφυλάξουν. Επίσης, ε, δεύτερη πυλώνας που μπορεί να είναι και συλλογική και υποχρεωτική να έχουν προτεραιότητα. Και στα εξωτικά συστήματα δεύτερου πυλώνα συνήθως συνδέονται με μεγάλες εταιρείες και μπορούν να χρηματοδοτηθούν και διακλαδικά, διατομεακά. Φυσικά θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα κάνουμε το καθήκον μας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεχνούμε και την ανάγκη ε, διαπαιδαγώγησης και των εθνικών μας κοινοβουλίων και των κυβερνήσεών μας. Γιατί δυστυχώς ε, έχουν εγκλωβιστεί σε παροχημένη συζήτηση και δεν θέλουν καθόλου να σκέφτεται τη πιθανότητα κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν. Ε, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις νέες ε, συνθήκες και να μην φοβούνται πια να ασχοληθούν με τα συνταξιοδοτικά. Έχει γίνει σαν η σύνταξη. Έχει επανέλθει η κυρία Γεζοβιέτσκα θα της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας για την έκθεση που περιλαμβάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση κατάστασης και περιγραφή των σημαντικών προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και τις ανάγκες μεταρρυθμίσεων των συνταξιδοτικών του συστημάτων. Πιστεύω ότι πολύ σωστά τονίζει η εισηγήτρια το γεγονός ότι αν θέλουμε καλές συντάξει θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και έγκυρη είσοδο στην αγορά εργασίας και παραμονή του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας. Μόνο έτσι θα υπάρχει δυνατότητα καλής προετοιμασίας και για την ε, εποχή της σύνταξης. Βέβαια λέμε ότι θα είναι δύσκολο στο μέλλον να χρηματοδοτήσουμε συντάξεις από τον κρατικό κορβανά και σήμερα πάνω από το 20% των νέων δεν μπορούν καν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και έτσι να προετοιμάσουν τη σύνταξή τους για αργότερα. Φυσικά και είμαι υπέρ των πρωτοβουλειών ε, για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των ενηλίκων άνω των 50 ή των 55 και βελτίωση των εργασιακών συνθήκων ε, για να επιτρέπουν την όσο δυνατόν πιο μακροχρόνια παραμονή και αποτελεσματική παραμονή στην αγορά εργασίας. Πολύ σωστά επίσης η εισηγήτρια μας επισημαίνει την ανάγκη σύνεση σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για, τις, ε, για, για τα επικουρικά προαιρετικά συστήματα συντάξεων και η αλλαγή της οδηγίας ίσως δημιουργήσει αύξηση του κόστους και αποτρέψει, αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις ε, ε, από προσφυγή σε τέτοια συστήματα προαιρετικά. Επίσης, διακόπτη η πρόεδρος. Δυστυχώς εξαντλήσετε το χρόνο σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Τελευταία πρόταση, παρακαλώ. Ολοκληρώστε αμέσως. Είναι αφισβήτητο ότι η οδηγία αυτή που αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι σημαντική για την ενίσχυση της κινητικότητας, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω λοιπόν την εισηγήτρια, αντί να αναφέρεται στους τρεις πυλώνες μόνο, να λέει για τι σύστημα πρόκειται. Αν πρόκειται για ε, δημόσιο σύστημα συντάξεων ή ιδιωτικό ή επιχειρησιακό. Γιατί ε, δεν υπάρχει κοινή συμφωνία για το πώς αντιμετωπίζονται οι πυλώνες και σε τι αντιστοιχούν οι πυλώνες. Ευχαριστώ. Σα δίνω το λόγο τώρα στην Κομισιόν. Μπορώ να σα δώσω μόνο τρία λεπτά. Ξέρω πω δεν αρκούν, αλλά έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη και πρέπει οπωσδήποτε να τα εξετάσουμε. Τρία, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την συγγήτρια για την γενική έγκριση των βασικών μας ε, με μηνυμάτων που έχουμε προτείνει στο Λευκό Βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι είμαστε στο ίδιο πνεύμα σε τόσο σημαντικά θέματα. Γιατί η δουλειά για περισσότερα χρόνια είναι βασική, ε, ο βασικός δρόμος για να εξασφαλίσουμε την συνταξιδοτική κάλυψη στο μέλλον και επίσης για τη δυνατότητα εργασίας των ε, ηλικιωμένων εργαζομένων και η απασχόληση των νέων δεν είναι αντιφατική στόχη. Όλα αυτά λοιπόν παραμένουν ε, ως πυρήνας της κατάλληλης σύνταξης στο μέλλον για να διαμπορέσουν οι πολίτες να εξοικονομήσουν σε συμπεπικουρικά δεξιδοτικά συστήματα. Ε, κατανοούμε τις ανησυχίες σας, κυρίως όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας IORP για τα συστήματα απασχόλησης, καθώς και τα σχόλιά σας για το Ευρωπαϊκό Συνταξιδοτικό Ταμείο για την έρευνα, για τους ερευνητές μάλλον. Ε, θα λαμβάνουμε υπόψη αυτά όλα, τις ανησυχίες σας και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Ναι, αλλά πρέπει να σας δώσουμε ναι, με το λόγο, αλλά πρέπει να απαντήσετε κιόλας. Η συγκίτρια σας ρώτησε γιατί εσείς σκοπεύετε κυρίως τους ε, ερευνητές. Να εντάξει, ε, μας είπατε απλά ότι θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Μα σας θέσαμε συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν δεν έχετε όμως ιδέες, αφήστε το, δεν πειράζει. Ειδικό καθεστώς για τους ερευνητές, λέτε, άρα κάτι πρέπει να έχετε υπόψη αυτή τη στιγμή η ιδέα αυτή είναι σε πιλωτικό στάδιο. Δεν, θέλουμε, δεν έχουμε δηλαδή τίποτα υποχρεωτικό ή πανευρωπαϊκό προσχέδιο. Είναι μια μικρή συμμαχία των προθήμων κάποιων πανεπιστημίων που γίνεται αυτή τη στιγμή με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το, κάποια, κάποια ταμεία έχουν δείξει ενδιαφέρον. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πόρα απέχουμε από οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα πανευρωπαϊκό ευρωπαϊκό σχέδιο. Μάλιστα. Ήδη κάπως μας τα συγκεκριμονοποιήσατε. Η συγγήτρια. Ναι, Πρόεδρε. Δεν νομίζω πως ένα ειδικό ταμείο για τους ερευνητέ θα λειτουργούσε. Έχω δει ερευνητέ, μάλλον ένα ερευνητή από τη Γαλλία ή την Γερμανία θέλει να πάει στην Ελλάδα, όπου ισχύουν τελείω διαφορετικοί μισθοί. Πώ αυτό το σωματώσετε σε ένα ενιαίο ταμείο, Περισσότερα προβλήματα μου φαίνεται θα, θα δημιουργήσουμε. Λοιπόν, αλληλεγγύη, ναι, αλληλεγγύη είναι και παραμένει σημαντική άσχετα από το ποιο σύστημα θα έχουμε. Όχι μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και στις γενναίες. Η φτώχεια, τα αξιοπρεπή εισοδήματα, το πρόβλημα όμως είναι ότι μόλις γίνονται περικοπές, τα πρώτα εισοδήματα που επηρεάζονται είναι αυτά των συνταξιούχων. Και Φαίνεται να γίνεται λόγος μόνο για προσαρμογή του ορίου συνταξιδότησης. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, ε, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος πάνω από τα 55 θα ήθελε να δουλέψει. Έχει απολυθεί και δεν μπορεί να ξαναβρει δουλειά. Ε, ας πούμε, στην ε, Ολλανδία το πρώτο που καταργήθηκε είναι αυτό το υποτιθέμενο ταμείο ζωτικ, ζωτικότητας, όπως λέγεται. Ε, τώρα, τα συνταξιδοτικά προγράμματα, ε, ε, τα επικουρικά. Λέει η Κομισιόν τα επικουρικά να έχουν κεφάλαιο εξ αρχής και να ενθαρρύνονται η ιδιωτική αποταμίευση. Μα εμείς όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, όσον αφορά συλλογικέ λύσει. Δεν πρόκειται για αλληλεγγύη ανάμεσα στι γενναίε, αλλά για συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και από τι δύο πλευρέ του κλάδου. Και έπειτα για τον κύριο Τεμπάκερ. Μιλούσε για ασφαλίσεις, ασφαλίσεις που έχουν πολλά κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν. Όμως οι επενδύσεις είναι διαφορετικά, ε, ε, διαφορετικές από, μάλλον οι ασφαλιστικές εταιρείε είναι διαφορετικές από τα εξαιρετικά ταμεία. Τα εξαιρετικά ταμεία σχετίζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και διαχειρίζονται τις εξοικονομήσεις τις αποταμιεύσεις των, των ε, συνταξιούχων. Μία ασφαλιστική εταιρεία όμως έχει εμπορικού στόχους. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά θα πρέπει να το δούμε ότι είναι διαφορετικές. Και έπειτα, τι πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση, να λάβουμε υπόψη στο πράσινο βιβλίο, δυνατότητα μεταφοράς και κινητικότητα. Αυτά όλα θα πρέπει να μεταφραστούν. Δεν μιλάω μόνο για κινητικότητα ανάμεσα στις χώρες, αλλά και μέσα σε ένα κράτος μέλος. Αν θέλουμε να έχουμε περισσότερη κινητικότητα, Εάν θέλουμε να έχουμε πέντε χρόνια παραπάνω, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί σε πέντε χρόνια μπορεί κανείς να μετακινηθεί. Και άρα οι, οι καταβολές θα χαθούν. Και αυτά είναι πολύ σαφή για τις γυναίκες που πολύ συχνά ζουν στη φτώχεια, διότι η σύνταξή τους είναι εξαιρετικά μικρή. Ε, αυτά είναι στην παράγραφο 13. Δεν θέλω τώρα να τριβήσω περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Εγώ να αναφέρω κάτι το οποίο δεν ανέφερε η Κομισιόν, ότι ξέρετε τι συμβαίνει για τη δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων στο Συμβούλιο οι δεδομένες της οικονομικής κατάστασης, της παρότρησης στην κινητικότητα, ε, όχι, όχι αναγκαστική κινητικότητα, αλλά λόγω κρίσης κινητικότητα. Δυνατότητα μεταφορές ε, συνταξιωτικών δικαιωμάτων ε, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Το συζητήσαμε από το 2009 για νέα νομική βάση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και επανεσύχθη η προηγούμενη πρόταση γιατί η Κομισιόν δεν έβαλε νέο θέμα στο επιτάπητος. Δουλεύουμε στο παλιό κείμενο με τη νέα νομική βάση όμως. Που είναι ακριβώς αυτό το σενάριο που είχαμε ζητήσει, προβλέψει το 2009. Επ' αυτής της βάσης ανοίγει η, κατάθε... κατάθεση τροπολογιών για τις 8 πρώτου 13 θα εξεταστεί το κείμενο στις 20 και 21 Ιανουαρίου, συμβαστικές 20 Μαρτίου, ψηφοφορία την επόμενη, ώστε να φτάσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Γυρνούμε πίσω στο χρόνο. Ο κ. Χάουιτ μπόρεσε να προσέλθει παρόλο που τον καθυστέρησε η κυκλοφορία. Ευχαριστώ τους Γερμινείς μας παρεχώρησαν 10 λεπτά. Θα χρειαστεί βεβαίως να είμαστε αυστηροί με την τήρηση του χρόνου. Εσείς κύριε Χάουιτ, σας παρακαλώ να μας παρουσιάσετε πολύ σύντομα τις τροπολογίες που έχουν κατατηθεί για τις δύο εκθέσεις σας. Η πρώτη έκθεση είναι εκεί όπου βρίσκεστε σε ενισχυμένη συνεργασία με την Νομική Επιτροπή για γνωμοδότηση και η δεύτερη έκθεσή σας εκείνη στην οποία έχετε πλήρω την ευθύνη. Και οι δύο εκθέσεις αναφέρονται στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων. Έχετε το λόγο αγαπητέ κύριε. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, αλλά κόπηκε το ρεύμα μέσα στο τούνελ ε, που βρίσκεται το τραμ. Έχουμε λοιπόν τώρα προδιαγραφές και άλλα και ευχαριστώ πολύ που έχω, μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω σύντομα τις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ ιδίως τους άλλους όπως ε, τον κύριο Μαν. Δεν μπορώ να σχολιάσω πλήρως τις δικές του τροπολογίες λόγω αγνίας των γερμανικών, αλλά ε, γνωρίζω που βρίσκεται και ελπίζω, το ίδιο και με την κυρία Φοντανιέ, διάβασα τα ισπανικά των, στα ισπανικά της τροπολογίας της και θα συνεργαστώ και μαζί τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω ότι θα επιτύχουμε σημαντική συνένεση στα πλαίσια της παρούσας επιτροφής. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μου έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες για τα θέματα αυτά και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία τους θα τα καταφέρουμε. Έχω καταθέσει ορισμένες εργατικές μετροπολογίες, όλες όμως περιλαμβάνονται στην επεξηγηματική δήλωση που έχει δημοσιευτεί ήδη. Δεν υπάρχουν λοιπόν εκπλήξεις έχω υποβάλει και ορισμένε αντικειμενικέ τροπολογίε σχετικά με τα παγκόσμια στάνταρτ και ε, των Ηνωμένων Εθνών για ε, επίσης των διεθνών το τυπο, οργανισμών τυποποίησης για την αεφόρο ανάπτυξη και του ΟΣΑ. Το κείμενό μου δεν θα είναι ακριβές 100% με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αν είναι δυνατόν να ε, συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή για την... Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια και για το ξεπέρασμα της κρίσης. Η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει και κείμενο για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες για τον τομέα ICT και υπάρχουν και ορισμένε τροπολογίε και δικέ μου και του Steven Hughes για τι συνθήκε απασχόληση. Προτείνω στόχο για τις νέες συμφωνίες πλαίσια και για τη λεγόμενη capacity building, προγράμματα δηλαδή δημιουργίας ε, capacity σε ορισμένες και σε τρίτες χώρες και πιστεύω ότι στη συνεργασία με τους συναδέλφους μου θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ ζητώ στις δικές μου τροπολογίες να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συμμετοχή και παγκόσμια και η Κομισιόν να δώσει το παράδειγμα. Τώρα σε ό,τι αφορά άλλα μέλη της Επιτροπής υποστηρίζω τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει ο κ. Μπουλόν, για κοινωνικούς δείκτες. Επιθυμώ να συζητήσω μαζί του τα λεγόμενα social labels. Εγώ διστάζω να υποστηρίξω την ιδέα αυτή, αλλά θέλω να συζητήσω μαζί του. Βρίσκω, έχω κατανόηση για τις ε, τροπολογίες της κ. Παπαδοπούλου και, και άλλων συναδέφων, τον του κ. Πουπάκη, επίσης για τις ε, μικρές επιχειρήσεις, τον κ. Τάκουλα, που νομίζω ότι όλες αυτές συμβιβάζονται με τις δικές μου τροπολογίες του ίδιου για θέματα ισότητας των φύλων. Είναι σημαντικό να μην επαναλαμβάνω τα πράγματα αυτά βέβαια σε όλες τις τροπολογίες και πιστεύω ότι θα μπορέσω να υποστηρίξω πολλές από τις τροπολογίες αυτές. Για τις συμβαστικές τροπολογίες μίλησα και με τον παλαιό μου φίλο και συνάδελφο Τόμας Μάν. Δεν συμφωνούμε βέβαια απολύτως, αλλά από την κοινότητα των επιχειρηματιών άκουσε ότι οι νέοι ορισμοί της Κομισιόν τους βρίσκουν σύμφωνους και αυτά που έχουν συμφωνήσει και στα Ηνωμένα Έθνη οι εργοδότες είναι κάτι που μπορεί να μας βρει και εδώ σύμφωνος. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του ή και της χώρας του, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό στα θέματα αυτά που τον ενδιαφέρουν, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε πλέον σε πολύ διαφορετικές θέσεις από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Και για παράδειγμα δική μου τροπολογία 20 για μια προσέγγιση ισορροπημένη και διαφοροποιημένη. Τώρα για ορισμένες... Για την ε, κυρία Μπερναμπέ, ε, ε, η Πρόεδρο, σας παρακαλώ ολοκληρώστε εδώ γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο. 20 δευτερόλεπτα για την οικονομική διαφάνεια. Ορισμένοι συνάδελφοί μου έχουν καταθέσει ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Εκεί θα χρειαστούμε γνωμοδότηση να στα εξετάσει και η κυρία Εσέ. Και Και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για την γνωμοδότηση και προς την άλλη επιτροπή. Μπουλάν πρώτα. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χόουιτ για την έκθεσή του και την γνωμοδότηση προς την ε, Νομική Επιτροπή. Πολύ καλές και οι δύο προσπάθειες. Για την γνωμοδότηση προς την Νομική Επιτροπή. Ε, θα πρέπει ε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη να είναι θέμα υποχρεωτικό και μάλιστα να περιληφθεί και ε, στα πανεπιστήμια ως πρόγραμμα σπουδών ε, και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θέλουμε μεγαλύτερη διάδοση αυτού του θέματος και να έχουμε ειδικευμένους οργανισμούς για να προσδιορίζονται οι κοινωνικές προδιαγραφές και κανόνες. Γιατί οι περιβαλλοντικοί κανόνες είναι πιο ποσοτικοποιήσιμοι, κάτι που δεν ισχύει για τους κοινωνικούς. Επίσης μια άλλη ιδέα ε, είναι με συγκεκριμένο σήμα να εντοπίζουμε τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων και βάλτιστων των πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων. Και με συγκεκριμένο σήμα ετικέτα της εταιρεία που χρησιμοποιεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να υποφεληθούν από την καλή εικόνα που δημιουργούν και προς τους καταναλωτές. Ελπίζω αυτή την πρόταση του ειδικού σήματο εταιρική κοινωνικής ευθύνης, ε, του κοινωνικού σήματο ουσιαστικά, να την ασθενιστεί ο εισηγητή. Αυτά είμαι σκιώδη εισηγητή τη ομάδα και είμαι στη διάθεση του εισηγητού για συμβαστικέ τροπολογίε. Ο Τόμας Μάν, ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίτσαρτ και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Γνωρίζει ότι ο εθελοντικό χαρακτήρα μπορεί να είναι εγγυημένο. Εσύ λε πάντοτε ότι οι επιχειρήσει κάνουν πολύ λίγα πράγματα και πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά τα πράγματα αυτά. Εγώ είπα ότι πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Οι καταστροφέ που, που, βλέπουμε τώρα στον εφαντουργικό τομέα ε, που έγινε στο Μπαγκλαντέ ή στο Πακιστάν. Αφόρητα πράγματα. Ο τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται του ανθρώπου εκεί και οι οποίοι εργάζονται υπό άθλιε συνθήκε δεν έχουν καμία σχέση βεβαίω με κοινωνικό προσανατολισμό. Αλλά πρέπει να διακρίνουμε το τι γίνεται στο CSR στις μικρέ και μεσέ επιχειρήσει με επιτυχία. Όπου δηλαδή ε, υπάρχει πραγματική ε, δέσμευση. Αν το ξεχωρίσουμε αυτό θα επιτύχουμε. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, για τι άθλιε συνθήκες των ανθρώπων που εργάζονται για να μπορούν να επιβιώσουν, αλλά αυτή πρέπει να είναι μια ξεχωριστή θέση. Γι' αυτό προσπάθησα εγώ να περάσω ένα στοιχείο διαφοροποίηση. να πούμε δηλαδή ε, ξεκάθαρη θέση για δέσμευση και αυτοδέσμευση και ξεχωριστά την, ε, τον, τον εθελοντικό χαρακτήρα του CSR. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, κάτι το οποίο θα με ικανοποιήσει πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφου που ήταν ε, πολύ αποτελεσματική στη χρήση του χρόνου. Θέλει ο συγκεκριτής ε, να δευτερολογήσει. Έφυγε ο κύριος Μπουλό. Πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε συμβαστικές τροπολογίες. Και σίγουρα ε, το θέμα της, του κοινωνικού σήματος ε, είναι σημαντικό. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με το, μεταξύ μας και ιδιαίτερα με τους και ηγητές. Πολύ ωραία. Οπότε... θα ψηφίσουμε τις διεκθέσεις της 14 Ιανουαρίου για να τις συζητήσουμε εγκαίρως και με την Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και ραντεβού στην επόμενη μας συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ. Ε, να είστε όσο δυνατόν περισσότεροι γίνεται. Ευχαριστώ.